Proszę Państwa. Otwieram dzisiejsze posiedzenie komisji. Bardzo Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο μας μάλλον μεταφέραμε από τη χτεσινή συνεδρίαση σε σχέση με τις ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα εργειακά προϊόντα και πρόθεσή τους στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. Επιλύθηκε το πρόβλημα που είχαμε με το Συμβούλιο και είχαμε αποφασίσει ότι θα συζητούσαμε αυτό το θέμα κατόπιν τροποποιήσεων το Σεπτέμβριο. Να το συζητήσει μόνιμη επιτροπή στο τέλη του Ιουλίου. Συζητήθηκε αυτό το θέμα και αποφασίστηκε ότι θα πάει στην επόμενη διαθέσιμη ολομέλεια της επόμενης θητείας. και είχαμε πει ότι θα το προσεγγίζαμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, σημαίνει ότι εγκρίνεται το εγγραφό αυτό ομόφωνα στην Επιτροπή μας. Υπάρχει κάποιος που να έχει αντίρρηση με αυτό. Αν όχι, μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτό το διορθωτικό και να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Η κυρία Χάσελκα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η διαφήμιση και η υπεροχή ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα πιστεύουμε ότι είναι κάτι περιττό μπορούν να το κάνουν αυτό οι παραγωγοί. Πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβα ένα σχόλιο κάνατε, όχι ότι είχατε κάποια αντίρρηση. Επομένως μπορούμε να δεχτούμε το διορθωτικό αυτό. Ευχαριστώ. συνέχεια περάσουμε σε ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό, όπως γνωρίζετε όλοι. Υπάρχει ένα εμπάρκο από τις 7 ε, Αυγούστου έναντι των ευρωπαϊκών προϊόντων που εισάγονται στη Ρωσία. Ο τομέα των απορροκυπευτικών έχει πληγεί ιδιαίτερα, όπως και ο γαλακτοκομικός τομέας, αλλά και ο τομέας του κρέατος. Πρόκειται για μια κατάσταση που πλήττει πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων την δική μου, που είναι η κυρία Προμηθεύτρια, χώρα Μήλων, στη Ρωσία. Και επομένως ε, χρειάζεται μια επίγουσα λύση η παραγωγή, έτσι ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν τη σοδιά τους. Είμαι βεβαισμένος ότι και εσείς συνάδελφοι έχετε παρόμοιες ανησυχίες που σας εκφράζουν η παραγωγή από διάφορους κλάδους. Επομένως, η διάσταση του προβλήματος αυτού είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Θα ήθελα και πάλι να καλωσορίσω τον κύριο Κόρτε από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη, ο οποίος ε, είναι αρμόδιος για τις γεωργικές αγορές και θα μας παρουσιάσει τα μέτρα που έχει θετήσει η Κομισιόν ώστε με αυτής της κατεπίγουσας διαδικασίας αναφερθεί επίση και στις τελευταίες αλλαγέ τάσεις τη αγορά και ποια είναι τα μέτρα που έχει προετοιμάσει η Κομισιόν. Παρακαλώ κύριε Κόρτε, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν ε, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα το πρωί να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας για την ρωσική απαγόρευση προϊόντων διατροφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Στην παρουσία μας καταρχήν να πω λίγα λόγια για τον αντίκτυπο της απαγόρευσης που είναι πολύ σοβαρός Δεύτερον, να παρουσιάσω την απάντηση της Κομισιόν μέχρι τώρα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα μέτρα που εξετάζουμε. Και τρίτον, να αναφερθώ στο ενημερωτικό σημείωμα που υιοθέτησε χθε Επιτροπό και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει διαβιβαστεί σε όλου σα μέσω τη Γραμματεία. Χθε ε, το Σώμα των Επιτρόπων ε, συναντήθηκε και συζήτησε αυτή την ε, απαγόρευση εισαγωγή σε ένα σημείο που παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Τσόλο, το οποίο τώρα έχει διατεθεί σε εσά αλλά και σε όλα τα κρατη Το πρώτο μου σημείο για τον αντίκτυπο τη απαγόρευση, όπω είπατε και εσεί πρόεδρε, η απαγόρευση εισαγωγή ε, που αποφασίστηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία στι 6 και 7 Αυγούστου έχει έναν ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Γεωργία όλα τα τρόφιμα και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα κρέματος ε, έχουν ε, υπαχθεί από τη μια μέρα στην άλλη σε αυτή την απαγόρευση και αυτό πιέζει πολύ έντονα τον γεωργικό τομέα και τον τομέα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να φερθώ σε δύο συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι η προσωρινή ελπίζουμε απώλεια μιας πολύ σημαντικής αγοράς στη Ρωσία είναι ο δεύτερος πελάτης μας ε, για αγροδιατροφικά προϊόντα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά μέσο όρο 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ εξάγονται στη Ρωσία κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη ε, και συγκεκριμένοι κλάδοι πλήττονται το 29% των εξαγωγών σε φρούτα και λαχανικά έχει σταματήσει το 33% των εξαγωγών τυριών και 28% του εξαγωγής βουτύρου. Αυτά είναι τα μερίδια των εξαγωγών. Αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία των εξαγωγών σε σχέση με την παραγωγή, η κατάσταση είναι διαφορετική ενώ το 29% ε, των ε, τροφίμων και λαχανικών απαγορεύεται ε, να ξεχθώ, αυτό αποτελεί μόνο το 1,7% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το τυρί είπα ότι πλήττει το 33% των εξαγωγών, αυτό αποτελεί το 2,7% της παραγωγής. Επομένως, ενώ είναι σοβαρός ο αντίκτυπος της απαγόρευσης, δεν θα πρέπει ούτε να υπερβάλλουμε σε σχέση με την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο ένα αρκετά περιορισμένο τμήμα της παραγωγής μας πλήττεται, όμως έχει χαθεί μια σημαντική εξαγωγική αγορά. Επίσης, ε, φυσικά θα έχουμε ως αποτέλεσμα υπερπροσφορά στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά τα προϊόντα πρέπει κάπου να καπάνε και αυτό είναι ένα δευτερογενές αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα λιλουχίας που προσπαθούμε να μετρήσουμε. Αυτό είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για τον τομέα των απορροκυπευτικών, ε, όπου ε, άρχισε η απαγόρευση στη μέση της ε, σεζόν της συγκομιδής. Κάπου πρέπει να πάνε τα προϊόντα λοιπόν και αυτή η κατάσταση έχει καθορίσει την απάντηση που έχει λάβει η Κομισιόν μέχρι τώρα. Και φυσικά θα ήθελα να πω από την αρχή ότι η αλληλεγγύη είναι κλειδί και το πιστεύει αυτό και ο Επίτροπο Τσόλο. Πρέπει να έχουμε μία μοναδική απάντηση, μία μοναδική απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην απαγόρευση και στην απειλή στου γεωργού μα. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει ένα ολοκλήρο οπλοστάσιο μέσων για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν είναι μια σοβαρή κατάσταση Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον στην εξωτερική μας επικοινωνία για να δείξουμε ότι είμαστε ενθεκτικοί και κατόπιν όσο είπαν και τα κράτη-μέλη το καλοκαίρι. Ε, μπορώ να πω ότι ήταν μετρημένα στην απάντησή τους και ήταν καλή η αντίδραση αυτή, τουλάχιστον γιατί δεν πρέπει να δώσουμε ένα επιπλέον δώρο στον κύριο Πούτιν, δηλαδή δείχνοντας ε, ότι υποχωρούμε και ότι παθαίνουμε πανικό. Τι έχει κάνει η Κομισιόν για να απαντήσει στην απαγόρευση αυτή της 6ης και 7ης Αυγούστου. Καταρχήν, οργανώσαμε εβδομαδιαίες συναντήσεις με τα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο στις χώρες τους και στους διάφορους κλάδους. Αυτές οι συναντήσεις βοήθησαν πολύ την Κομισιόν γιατί μας έδωσαν πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία και συνεισφορά που τη χρειαζόμαστε προκειμένου να λάβουμε μέτρα που πραγματικά βοηθούν. Επίσης, ε, Εντείναμε την παρακολούθηση των ιδιωτικών αγορών ε, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και βάλαμε αυτά τα στοιχεία στις ιστοσελίδες μας έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους. Και κάθε πληροφορία που έχουμε είναι πραγματικά διαθέσιμη σε όποιον θέλει να τη δει. Και πήραμε μέτρα. Αυτό είναι το τρίτο σημείο. Κινηθήκαμε γρήγορα από το σημείο που υιοθέτησε η Κομισιόν θα δείτε μια προσέγγιση σε τρία στάδια. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο κατεπήγον βήμα ήταν η σταθεροποίηση της αγοράς ε, για τα αναλώσιμα, κυρίως για τα φρούτα και τα λαχανικά. Αυτή η απόφαση λήφθηκε τον Αύγουστο. Το δεύτερο στάδιο είναι μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς για τα γαλακτοκομικά και τέσσερα μέτρα θα ληφθούν σήμερα από την Κομισιόν. Και τρίτον, παρακολουθούμε και αναλύουμε τι υπόλοιπε αγορές που έχουν πληγεί και αυτό αφορά κυρίω την αγορά του κρέατος και εξετάζουμε νέα μέτρα. Καταρχήν λοιπόν φρούτα και λαχανικά, δεύτερον γαλακτοκομικό τομέα και τρίτον τομέα του κρέατος. Για το πρώτο και για το δεύτερο τομέα και για τα γαλακτοκομικά έχουμε πάρει μέτρα και για το τρίτο το εξετάζουμε, παρακολουθούμε τι αγορέ και συζητούμε και στο και με τα κρατημέλη αν χρειάζονται μέτρα. Ο Επίτροπος Τσόλος από την αρχή ξεκαθάρισε ότι ήθελε να κινηθεί γρήγορα και ότι πίστευε ότι είναι καλύτερο να λάβουμε γρήγορες αποφάσεις ακόμη και αν δεν έχουμε πάντοτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεσή μας για να δικαιολογήσουμε το ένα ή το άλλο μέτρο στην ε, τελευταία του λεπτομέρεια. Για να είμαι ειλικρινής, μερικές φορές λαμβάνουμε μέτρα σε κάποια βάση που δεν είναι 100% αξιόπιστη, αλλά είναι καλύτερο από το να περιμένουμε μέχρι να ξέρουμε, γιατί τότε θα είναι υψηλότερο το κόστος. Ε, φυσικά το να λαμβάνουμε γρήγορα μέτρα, ελπίζουμε ότι έχει καλό ψυχολογικό και πολιτικό αντίκτυπο, δηλαδή όλοι γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν είναι εδώ και θα έρθει να βοηθήσει. Τώρα, πολύ γρήγορα να πω δύο λόγια για τα μέτρα που έχουμε λάβει για τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα δείτε από το σημείωμα, θα δείτε και στον τύπο της 11 Αυγούστου, υιοθετήσαμε ένα μέτρο να δώσουμε επιδοτήσεις για την απόσυρση από την αγορά για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και στις 18 Αυγούστου ανακοινήσαμε ένα επιπλέον μέτρο που καλύπτει 13 κατηγορίες φρούτων και λαχανικών που έχουν ιδιαίτερα πληγή από την απαγόρευση. Και τα δύο μέτρα δεν είναι τα ίδια. Έχουν κάποιες διαφορές, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε τώρα εδώ σε λεπτομέρειες. Όμως και τα δύο μέτρα προβλέπουν χρηματοοικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόσυρση φρούτων και λαχανικών με διάφορα μέσα για ελεύθερο προορισμό, όπως καλείται, δηλαδή για φιλοθροπικούς σκοπούς, αλλά ε, και για πρώιμο, πρώιμη σοδιά ή για καταστροφή. Ελπίζουμε ότι η καταστροφή είναι το έσχατο μέσο το έσχατο μέτρο που λαμβάνεται. Αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται και οι οργανώσεις παραγωγών και τα κράτη-μέλη και οι γεωργοί τα χρησιμοποιούν. Φυσικά σήμερα δεν είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσω ιδιαίτερε λεπτομέρειες για την πρόσληψη αυτών των μέτρων. Εμείς ε, φυσικά θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα κρατη και πώς οι γεωργοί αντιδρούν σε ε, αυτά τα μέτρα στήριξης, τα χρησιμοποιούν και σε ποιο βαθμό. Οι πρώτες κοινοποιήσεις θα έλθουν στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη αυτή την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα για την άμεση πρόσληψη αυτών των μέτρων. Τώρα πάμε στο γαλακτοκομικό τομέα, όπου θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Το νούμερα μας δείχνουν ότι είχαμε μεγάλη έκθεση στις ε, ρωσικές αγορές και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κακή σε ορισμένες χώρες ο αντίκτυπο τη απαγόρευση στα γαλακτοκομικά είναι αρκετά άνισος και θέλω να αναφέρω τις χώρες, κάποιες χώρες όπως Φιλανδία, Λιθουανία, Λετωνία, που πάνω από 90% εξαρτώνται από τη ρωσική αγορά για τις εξαγωγέ γαλακτοκομικών, αλλά και κάτω χώρες ω μεγάλο παραγωγό. η Γερμανία και η Πολωνία εξάγουν σημαντικέ ποσότητε στη Ρωσία. Εδώ η απαγόρευση ήδη συνεισφέρει σε μείωση, ε, σε πίεση των τιμών προς τα κάτω mm. στις αγορές. Ε, οι τιμές των γαλακτικών ήταν ε, ιδιαίτερα ψηλές τα τελευταία έτη. Έτσι λοιπόν τώρα από ένα πολύ ψηλό επίπεδο πηγαίνουμε προς τα κάτω. Και δεν είμαστε κοντά στο επίπεδο του δικτύου ασφαλείας που υπάρχει για να υπάρξει δημόσια παρέμβαση, εκτός ε, ίσως από αυτές τις χώρες της Βαλτικής που ανέφερα, αλλά δεν ε, έχουμε αγοράσει καθόλου βούτυρο ή γάλα σε σκόνη υπό το δημόσιο καθεστώς παρέμβασης. Μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον. Επίσης έχουμε καλέσει και μία πρώιμη συνάντηση του παρατηρητηρίου για το γάλα για να έχουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την αγορά. Τι κάναμε λοιπόν μέχρι τώρα για αυτούς. Τέσσερα μέτρα έχουν ληφθεί. Σήμερα η ιδιωτική αποθεματοποίηση ξεκίνησε για το βούτυρο και για το γάλα σε σκόνη, αποβυτρωμένο σε άλλο σε σκόνη και επίσης για το τυρί. Το τυρί που θα εξαγόταν στη Ρωσία. Και επίσης ο Επιτρόπος αποφάσισε σήμερα να διευρύνει την περίοδο κατά την οποία είναι ανοιχτέ οι δημόσιες παρεμβάσεις από τις 30 ε, Σεπτεμβρίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου. Και το τέλη Σεπτεμβρίου, στο μετά η δημόσια παρέμβαση και θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τελικά θα είμαστε εδώ για στήριξη μέχρι το τέλη του έτους, αν χρειαστεί. Αν και τίποτα δεν έχει αγοραστεί υπό τη δημόσια παρέμβαση μέχρι τώρα, πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο ψυχολογικά και πολιτικά βοηθά, γιατί βοηθά για να μπει ένα κατώτατο όριο στην αγορά. Τώρα για την αγορά κρέατο, τα πουλερικά, το χοιρινό κρέας και το βόλιο κρέας δεν έχουν ληφθεί μέτρα μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποφασίσουμε τίποτα, αυτό το ξεκαθαρίζω. Ο Επίτροπος Τσόλος είπε επανειλημμένα ότι είναι έτοιμο να μέτρα αν χρειαστεί, αλλά προς στιγμή δεν χρειάζεται, βλέπουμε ανάγκη να δράσουμε γρήγορα για την αγορά των πουλερικών. Έχει πολύ λίγο ε, ουσιαστικά επηρεαστεί, ε, εκτίθεται στη ρωσική αγορά, το 6% μόνο πηγαίνει στις αγορές, δηλαδή λιγότερο από το 1% της ε, κοινοτικής παραγωγής. Ξέρετε, είναι ευέλικτη η αγορά των πουλερικών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να αντιδράσει γρήγορα και να βρει μια άλλη διέξοδο. Αν χρειαστεί φυσικά να δράσουμε, θα το ξανακάνουμε. Το χοιρινό κρέας. Βρίσκεται σε μια περίεργη θέση ο κλάδος αυτός. Γιατί δεν υπήρχε μια απαγόρευση για το χοιρινό κρέας στη Ρωσία από νωρίτερα φέτος η Ρωσία είχε προβεί σε δικαιολόγητη απαγόρευση γιατί είχαμε κάποιες ε, περιπτώσεις ξεσόνοντος αφρικανικής πανόλης των χείρων. Έτσι λοιπόν ε, δεν προστίθεται τώρα τίποτα καινούριο για αυτό τον κλάδο, για αυτό τον τομέα. Παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά τις αγορές και αν χρειαστεί θα λάβουμε μέτρα και κατόπιν έχουμε το βόλιο κρέας τα γεγονότα είναι τα εξή. Είναι η ο πρώτος προορισμός η Ρωσία. Το 25% των εξαγωγών μας πήγαν στη Ρωσία. Τώρα, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε εναλλακτικέ διεξόδου αγορών. Δεν βλέπουμε ακόμη άμεσο αντίκτυπο στι τιμέ στον ε, τομέα αυτό. Η διαλογική ισχύ. Όταν μας ειδοποιήσουν τα κράτη-μέλη, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση. Τώρα θέλω να αναφέρω πολύ γρήγορα, γιατί ήδη έχω μακρηγορήσει. Να ευχαριστήσω την προσοχή σας σε μια σειρά άλλων μέτρων που θα μπορούσαν να ενδυνάμει να ληφθούν είτε από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα κράτη-μέλη και από τις επιχειρήσεις. Έχουμε και άλλα μέτρα στο πλωστασιό μας, ε, όπως σας είπα, όχι μόνο Το πρώτο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή τι θα κάνουμε στι εξωτερικέ μα αγορέ. Ελπίζουμε ότι θα έρθει σύντομα η απαγόρευση, αλλά ελπίζω ότι πολλοί επιχειρηματίε ε, πιστεύουν, πολλοί οικονομικοί φορείς πιστεύουν ότι δεν είναι αξιόπιστος εταίρο η Ρωσία. Έτσι λοιπόν πολλοί θα εξετάσουν θα προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτικέ αγορέ. Τι μπορούμε να κάνουμε να του βοηθήσουμε. Το πρώτο συμφέρον που έχουμε και προσπαθούμε τώρα να το εφαρμόσουμε για να άρουμε πολλά από τα εφιστάμενα εμπόδια στο εμπόριο που μας σταματούν από το να εξάγουμε αγκαθά ακόμη και σε τέρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, την Τουρκία ή άλλες χώρες. Έχουμε ακόμη πάρα πολλούς περιορισμούς υγειονομικούς και φυτογειονομικούς και έτσι είναι αδύνατο να εξάγουμε ε, φρέσκα προϊόντα σε αυτές τις χώρες. Θέλουμε λοιπόν να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Επίσης μέτρα προώθησης έχει γίνει μια ανακοίνωση, χτες ήδη έγινε από την Κομισιόν, θα διατεθούν περισσότερα χρήματα για μέτρα πρόθεσης σε τρίτες ε, αγορές, για να βρούμε νέες αγορές συνολεκτικές στη Ρωσία. Θέλω να αναφέρω και την κατανάλωση μέσω των προγραμμάτων για τη διανομή φρούτων και γάλακτος στα σχολεία. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν τη χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων. Θα θυμάστε ότι η Κομισιόν πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα για τη διανομή φρούτων και γάλακτος και συζητείται και εδώ και στο Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι αν επιταχύνουμε την διαδικασία θέτησης αυτής της πρότασης θα βοηθούσε. Γιατί αυτός ο νέος κανονισμός θα καθιστούσε ακόμη πιο εύκολα για τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την κατανάλωση γάλακτος και φρούτων και λαχανικών στα σχολεία. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα για τη διανομή τροφίμων στους απόρους, που έχουν τα κρατημέλη, από την αγροτική ανάπτυξη, από τα προγράμματα αγροτική ανάπτυξη που υιοθετήθηκαν πέρσι. Υπάρχει και μια σειρά μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη. Θέλω να τονίσω ένα, η σταθεροποίηση, το μέσο σταθεροποίηση του εισοδήματο που προβλέπεται ω επιλογή για τα κράτη-μέλη ως οψιόν. Αυτοί θα αποφασίσουν αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Δεν τη λαμβάνει αυτή την απόφαση Κομισιόν, αλλά τα κράτη-μέλη. Για να δούμε αυτό το μέσο. Φαίνεται ότι έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα όπως η απαγόρευση από τη Ρωσία. Θα επιτρέψει στους γεωργούς που έχουν ιδιαίτερα πληγή από την απαγόρευση να αποζημιωθούν. Mm. Όμως και πάλι την απόφαση αυτή πρέπει να αντιλάβουν τα κράτη-μέλη. Και τέλος, θέλω να φέρω την κρατική ενίσχυση όπου οι κανόνες επιτρέπουν κάποια ευελιξία για τα κρατη για να βοηθήσουν κλάδους και μονομενούς γεωργούς που έχουν ιδιαίτερα πληγή από αυτή την απαγόρευση. Βέβαια υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε κατάσταση να ανταγωνίζονται μεταξύ τους τα κράτη-μέλη κρατικές ενισχύσεις. Δεν θέλω να πω αυτό αλλά θα δείτε και ένα ενημερωτικό σημείωμα ότι υπάρχουν επιλογές, δυνατότητες, στις οποίες μπορούν να προσφύγουν στα κράτη-μέλη και θα συζητήσουμε μονομένες περιπτώσεις μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες για τη συζήτηση. Φυσικά πολλά ακόμη μπορούν να υποθούν. Η τελική Προεδρία του Συμβουλίου έχει καλέσει και μία έκτακτη συνάντηση των Υπουργών αύριο και ε, η Κομισιόν νομίζω θα παρουσιάσει τέτοια σημεία που σας παρουσιάζω και εγώ τώρα εδώ. Φυσικά, εμείς θέλουμε να συνεχιστεί περαιτέρω η συζήτηση και θέλουμε να έχουμε και την υποστήριξή σας. ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν το Σάββατο περιλαμβάνουν μία σειρά φράσεων για τις απαγόρευσεις και θα ήταν καλό αν και από την πλευρά του Κοινοβουλίου υπήρξε υποστήριξη, υπήρχε υποστήριξη για την Κομισιόν. Και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και να σας πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υποτιμούμε τις συνέπειες, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα αποφύγουμε και τον πανικό και θα ξεκινήσουμε από μια ισχυρή βάση. Και είναι η αγροτική πολιτική, όπως την μεταρρυθμίσατε και εσείς πέρσι, περιλαμβάνει μια σειρά χρήσιμων μέσων και δεν θα πρέπει να διστάσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε όλη την υποστήριξή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Ο κύριος Γλέζος έχει πρώτο το λόγο. Σας υπενθυμίζω ότι έχουν εγγραφεί 30 ομιλητές, οπότε ο, ο καθένας έχει ένα λεπτό. Μικρόφωνο στον ομιλητή παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση την οποία πρέπει να δούμε με πλήρη αντικειμενικότητα. Έχω μπροστά μου το κείμενο που παρουσίασε η Κομισιόν και ξεκινάει από το γεγονός ότι η Ρωσία επέβαλε αυτές τις ε, κυρώσεις. Αγνοεί ότι πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η Ατλαντική Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις και ακολούθησαν οι κυρώσεις από την άλλη πλευρά. Δηλαδή στην ουσία υποταχθήκαμε σε αυτό που έχω τονίσει και άλλες φορές στο εμπορικό ΝΑΤΟ. Σήμερα βλέπουμε και είμαστε μάρτυρες μιας κοκορομαχίας ανάμεσα στην Ατλαντική Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ρωσία. Ποιος εποφελείται από αυτή την κοκορομαχία μόνο οι έμποροι των όπλων οι οποίοι θα κερδίζουν από την πώληση των όπλων και είναι σε βάρος των λαών η κινητοποίηση του, του Ατλαντικού στρατού και ρωτάω ποιος πληρώνει τα έξοδα της κίνησης της διαδρομής του Ατλαντικού στρατού από τη βάση του έως την Ουκρανία. Την, πληρώνει, την πληρώνουν οι λαοί και οι λαοί είναι υποχρεωμένοι να υποστούν όλο αυτό το βάρος. Πέρα όμως από αυτό και πολύ μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι δημιουργείται ένα μίσος μεταξύ των λαών, μεταξύ των εθνών και είμαστε υπεύθυνοι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση εάν υποστηρίζουμε αυτού του είδους την πολιτική. Δεν επιτρέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να είναι παράγοντας ειρήνης μεταξύ των λαών που πρέπει να παίξει ένα ρόλο πρωταρχικό σε όλη αυτή την ιστορία να βοηθάει στην ανάπτυξη ενός μίσους μεταξύ των λαών. Άλλη μια φορά τονίζω ότι για την Ελλάδα ειδικά Έχουμε υποστεί τα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέλει την Ελλάδα θέρετρο. Τη θέλει ένα τεράστιο ξενοδοχείο και όχι να αναπτύξει την αγροτική της οικονομία και όλα τα μέτρα που πήρε ως τώρα ήταν εναντίον της ανάπτυξης αγροτικής οικονομίας. Bardzo dziękuję. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο ομιλίας δύο λεπτών, ο κύριος Μελό. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ γρήγορα. Οι πληροφορίες μας ε, παρουσιάστηκαν αναφέρουν γενικά τον αντίκτυπο για την Ευρώπη όμως δεν είναι ίδιος ο αντίκτυπος από χώρα σε χώρα. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, μια αξιολόγηση μας δείχνει ότι αυτό μας κόστησε 9 εκατομμύρια ευρώ για την ε, οικονομία. Εμείς έχουμε θυγεί ιδιαίτερα στον τομέα του χοιρινού κρέατος και στον τομέα των φρούτων και αυτό μας κόστησε 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό το σημείωμα που μας μοιράστηκε. Θέλω μία διευκρίνηση σε ορισμένα στοιχεία. Αναφέρεται σε αυτό το σημείωμα ότι μεταξύ των μέτρων έχουμε άμεσες αποζημιώσεις σε γεωργούς τους πιο πληγέντες τομείς. Όμως, μετά λέει, ανάλογα με την κλίμακα αυτού του μέτρου μπορεί να υπάρχει μία μείωση των άμεσων πληρωμών που σήμερα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους γεωργούς. Εγώ θα ήθελα να ξέρω σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Λοιπόν, για τη μείωση αυτών των άμεσων πληρωμών, εγώ θα ήθελα να ξέρω, προβλέπετε κάποια μέτρα για το άνοιγμα των ε, αγορών για να έρθουν κάποια εμπόδια στις εξαγωγές και αν λέγεται κάτι για αυτό ε, την αυστηρή έκφραση που λέει ότι μπορούν να ε, δοθούν αποζημιώσεις αν υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, αιτιολογείτε τώρα στην τρέχουσα περίπτωση αυτή η φράση έκτακτες περιστάσεις. Ε, Ευχαριστώ κύριο Χαϊτούμα. Όπως ε, ακούσαμε, η Ευρώπη είναι υποπίεση τώρα. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια, ε, τώρα ε, επιβάλλει μια μεγάλη εισφορά 400 εκατομμύρια, τα οποία θα αυξηθούν του χρόνου. Μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να τροποποιήσει τις ποσοστώσεις και να βγάλει την πίεση από αυτή την ε, υπερισφορά. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εδώ δεν είναι οι κατάλληλες. Παρ' όλα αυτά το μέτρο είναι καλό αφού τα χρήματα θα πάνε απευθείας στους αγρότες. Και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν πότε θα προβούν στην προσαρμογή αυτού του μέτρου. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικά ερωτήματα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Καταρχήν, δόθηκαν 127 εκατομμύρια για τα φρούτα και λαχανικά. Εγώ ζητώ περισσότερα. 125 εκατομμύρια δεν αρκούν ούτε μπορούν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Αυτά τα 125 εκατομμύρια δεν θα μπορούσαν να αυξηθούν και από άλλα ταμεία. Πόσο. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι έγινε από την κρίση του 11. Τότε η Κομισιόν είχε διαθέσει περισσότερα χρήματα. Γιατί στην τωρινή κρίση δεν κάνει το ίδιο. Θεωρεί μήπως η Κομισιόν ότι αυτή η κρίση είναι λιγότερο σημαντική Είχαμε μιλήσει για συνολική αποζημίωση της τιμής παρέμβασης και τώρα δεν εφαρμόζεται αυτό. Έχει την πρόθεση η Κομισιόν να καθορίσει καμία task force για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα των αγορών. Τι πρόοδους μπορούμε να πετύχουμε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Ευχαριστώ. Κανιέτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι γεωργοί της Λετωνίας εκπροσωπούν πάνω από 30% του δυναμικού μας και οι γαλακτοκομικές τιμές έχουν πέσει κατά 30% στη Λετωνία. 19 λεπτά το λίτρο, χαμηλότερο από το κόστος παραγωγής δηλαδή. Τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Κομισιόν είναι πραγματικά, αλλά ας δούμε ποιες είναι οι ποσοστώσεις των γαλακτοκομικών. 91,1% καλύπτουν για μας και δεν είναι σωστό στα πλαίσια αυτής της κρίσης να τιμωρήσουμε έτσι, να ζημιώσουμε τους γαλακτοπαραγωγούς. Προβλέπεται την άνοιξη του 2015 να καταργηθούν αυτές οι κυρώσεις και οι ποσοστώσεις γιατί έτσι, έτσι θα βελτιωνόταν η κατάσταση για τους παραγωγούς της Ανατολικής Ευρώπης αλλά μέχρι τώρα το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας δεν υποστηρίζει κανένα μέτρο τώρα. Πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη και ευελιξία για να επιτευχθεί ένα συμβιβασμός για τις κυρώσεις για το γάλα. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι και πολιτικό. Και μία φράση ακόμη, να μην νομίζετε ότι θα επιστρέψουν οι ρωσικές αγορές αν δεν υπάρξουν γεωπολιτικές αλλαγές που δεν θα δεχτεί ο Πούτιν. Ταντέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από ένα χρόνο έχει που όταν καθορίσαμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πολλοί ήθελα να μιλήσουμε και για την κρίση, αλλά δεν μάντευαν ποια κρίση θα ήταν αυτή. Είναι δυστυχώς διπλωματική η κρίση και είναι κρίμα που μόνο για τη γεωργία επιβάλλονται μέτρα. Θα ήθελα η Κομισιόν να μας υπενθυμίσει ποιο ήταν το αποτέλεσμα των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης στον πρώτο πυλώνα. Ανάλογα με τα ποσά θα μπορούσε να υπάρξει μείωση των επιχορηγήσεων ανά εκτάριο από του χρόνου. Άρα είναι απόλυτα απαραίτητο να σκεφτούμε να, ε, να λάβει περισσότερο υπόψη του προπολογισμό την αγροτική πολιτική που είναι ακόμη πολύ σημαντική. Ευχαριστώ κύριο Σράουπ, Παρακαλώ. Ε, ε, ε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα μέτρα για το γαλακτοκομικό τομέα που έχουν παρουσιαστεί δεν θα αρκέσουν αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα της κρίσης σε κάποιες χώρες, Φιλανδία, Λιθουανία κτλ. Φαίνονται να έχουν καταστροφικό σενάρια. Η Πορτογαλία βρίσκεται από την άλλη πλευρά της Ευρώπης, όμως ε, φυσικά και αυτή θα πληγεί στο γαλακτοκομικό τομέα. Εγώ προέρχομαι από τις Ασόρες, όπου η παραγωγή του γαλακτός αποτελεί το 3% της εθνικής παραγωγής. Η ευρωπαϊκή αγορά ε, θα πλημμυριστεί από γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν θα βρίσκουν διέξοδο και αυτό θα έχει άμεση συνέπεια ε, στους γεωργούς. Πέρα από τα μέτρα παρέμβασης που είναι επιτάπητος ε, δεν αρκούν για λόγους που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά και μεταξύ των οποίων η τιμή των 21 cents ε, ανά λίτρο που δεν φτάνει να καλύψει το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία δεν έχει την οικονομική ικανότητα για να θετήσει μέτρα κρατικών ενισχύσεων και θέλουμε μια ευρωπαϊκή λύση. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και προληπτικά. Είμαι σίγουρος ότι οι Πορτογάλοι κυβερνώντες θα θέσουν αυτό το θέμα στο Συμβούλιο που θα λάβει η χώρα αύριο. Εμείς δεν πρέπει φυσικά ε, να ε, ζητούμε πάντοτε από το Συμβούλιο να εξετάζει τα θέματα αυτά και να λαμβάνει συνεπή δράση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. za ublažavanje štete embarga e, οι κυρώσεις της Ρωσίας βλάπτουν την Ένωση. Εδώ και 15 μέρες το είχα ξαναπεί ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους γαλακτοπαραγωγούς και τους παραγωγούς μανδαρινίων. Στην Κροατία λόγω των ρωσικών κυρώσεων θα σημειωθούν απόλυες 25 εκατομμυρίων δολαρίων ο γαλακτοκομικός τομέας για μας, καθώς και τα μανταρίνια, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Η Κροατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εδώ και λίγο καιρό, αλλά γίνεται και θύμα των μέτρων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη. Έχω ξαναπεί στην Επιτροπή μας το έχω ξαναπεί και έχω ζητήσει επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη διανομή γάλακτος και φρούτων στα σχολεία. Αλλιώς θα πρόκειται στην ουσία για άνηση μεταχείριση. Σέντρα. Καταρχήν, να πω ότι εμείς οι Γεωργοί είμαστε θύματα μιας πολιτικής απόφασης που έλαβαν ε, οι κυβερνώντες μας ε, και έχουν την ευθύνη. Επίσης, ε, θέλω να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο της Κομισιόν και να του πω ότι είναι πολύ εύκολο να είναι κανείς γενναίος όταν αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή και η αξιοπρέπεια των γεωργών της Ευρώπης. Αν φυσικά διακυβευόταν ο δικό σα μισθών και ο μισθός όλων όσων πήρε αυτή την απόφαση, μάλλον δεν θα είχαμε καταλήξει εδώ. Σε σχέση τώρα με τα μέτρα που παρουσιάζετε εσείς, θα ήθελα να πω διάφορα. Καταρχήν, εσείς ε, αναφέρεστε σε κάποια μέτρα τα οποία είναι πολύ βραχυπρόθεσμα μέχρι τα τέλη του έτους είπατε για τα γαλακτοκομικά ή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για τα προκυπτευτικά και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία λύση μέχρι τότε. Θα έπρεπε λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς θα κάνετε από εκεί και πέρα. Δεύτερον, Μπαίνοντα τώρα στις λεπτομέρειες, ε, μας εκπλήσει που για το τομέα του κρέτους δεν υπήρχε κανένα μέτρο μέχρι τώρα, τον ξέρετε ότι πραγματικά πλήττεται. Δεύτερον, σε σχέση με το γαλοκτοκομικό τομέα, όπως ε, λέμε στη χώρα μου, ε, ε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της απόφασης πήρατε εσεί να καταργηθούν οι ποσοστώσεις και να υπάρχει απελευθέρωση και τώρα μας εκπλήσει που δεν υπάρχει κανένα μέτρο για να προσαρμοστεί η προσφορά στη ζήτηση. Επίσης, το ε, να προσαρμόζετε, ή, να προσαρμόζετε τιμές για κάθε ένα από τα προϊόντα, να μας λέτε κάτι τέτοιο, είναι γελίο. Τώρα, αν μιλήσουμε για τα απορροκυπευτικά, να σας πω ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει διαφορά διαφοροποίηση μεταξύ των ανθρώπων που είναι σε οργανώσει παραγωγών και των ανεξάρτητων γεωργών. Νομίζω ότι έχουμε την ελευθερία να είμαστε να μην είμαστε οργανωμένοι και κάτι τέτοιο πλήττει όλους τους γεωργούς, έτσι λοιπόν σε όλους πρέπει να δίνονται οι ενισχύσεις και η βοήθεια. Και κάτι τελευταίο, υπάρχουν προϊόντα που πλήττονται αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα μέτρα. Παρακαλώ, δεν θέλω να αναγκαστώ να σας κλείσω το μικρόφωνο. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι αγρότες είναι τα πρώτα θύματα της σύγκρουσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Οι Σλοβαίνοι παραγωγοί έχουν προβλήματα στον τομέα των φρούτων και φοβούμεθα ότι θα πληγεί και ο τομέας του γάλακτος και του κρέατος που είναι πιο σημαντική στη Σλοβενία. Υποστηρίζουμε τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε για την ταχεία δράση και στηρίζουμε τα μέτρα πρόθεσης γάλακτος και φρούτων στα σχολεία. Φοβούμεθα ότι ε, τα άλλα μέτρα όπως πρόρος, τρίγος, ε, καταστροφή των προϊόντων δεν είναι ικανοποιητικά. Εμείς θέλουμε εντονότερη πρόθεση των προϊόντων και τα μέτρα αυτά που έγιναν δεκτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την πληροφόρηση του. Βλέπουμε ότι η Κομισιόν κατανοεί την κατάσταση και οι επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης. Όμως τα μέτρα που προτείνει ακόμη και αν για ορισμένες χώρες θα δημιουργήσουν σταθεροποίηση, για άλλες όπως τις Βαλτικές χώρες ή τη Φιλανδία, τα μέτρα αυτά θα, είναι, θα αποδειχθούν ανεπαρκή. Θέλουμε πρόσθετα εναλλακτικά μέτρα, ιδιαίτερα για τους πιο ευαίσθητους τομείς που πλήττονται όχι μόνο από τα ρωσικά μέτρα αλλά και από τον αυθόδη πυρετό των χείρων. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν χωριστά πρόσθετα μέτρα για τις χώρες που πλήττονται από αυτή την κατάσταση. Όταν μειώνεται η παραγωγή κατά 20-30% υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αύξησης της ανεργίας και οι γεωργοί καθώς και οι βουλευτές των βαλτικών χωρών μαζί έχουν απευθυνθεί στην Κομισιόν και σε άλλα όργανα με το αίτημα αυτό πρόσθετων μέτρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Η κυρία Ντότζ. Ο Η Κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Ας δούμε κάποια μέτρα παρέμβασης που αναφέρατε. Η ιδιωτική αποθεματοποίηση και ενίσχυση εκεί είναι ε, προσδεκτή και η επέκταση. Δημόσια αποθεματοποίηση ε, επεκτείνεται την περίοδό της αλλά δεν εκπλήσει ότι δεν χρησιμοποιείται αυτή στη Βόρεια Ιρλανδία στην εκλογική μου περιφέρεια το κόστος παραγωγής είναι περίπου 25-26 πένες το λίτρο ότι η τιμή παρέμβασης ε, είναι τρομερά χαμηλή και έχουμε και με παρατεταμένη περίοδο τώρα πολύ χαμηλών τιμών μέχρι να έχουμε την τιμή της παρέμβασης θα έχουμε το γαλακτοκομικό τομέα μέσα στην κρίση όπως συνέβη το 2008 και 2009. Είναι καιρός να εξετάσουμε την ιδέα επανεισαγωγής επιστροφών κατά τις εξαγωγές για να μπορέσουμε να έχουμε μία ε, ε, διέξοδο στην αγορά. Το κάνουμε, τα κάνουμε αυτά δε ε, μία περίοδο όπου θα τελειώσουν του χρόνου οι ποσοστώσεις. Νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση για το συγκεκριμένο αυτό θέμα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε σταδιακά να χαλαρώσουμε τους περιορισμούς των ποσοστώσεων και όχι να τις καταργήσουμε άπαξ ή διαπαντός. Βόρεια Ιρλανδία επηρεάζεται πάρα πολύ ε, λόγω των εξαγωγών βουτύρου και τυριού στη Ρωσία και πρέπει το Ταμείο για την Κρίση να το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε λίστα ο μεγάλο μας πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριος Χάουσλιν. Ευχαριστώ. Χρειάζονται αλληλεγγύη οι αγρότες, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιοι έχουν πληγεί ε, περισσότερο από τους άλλους, όπως οι χώρες της Βαλτικής. Όμως ένα βασικό ερώτημα είναι αν ο πολιτικός μας προσανατολισμός στις εξαγωγές ε, και στο γάλα κυρίως ε, ήταν σωστό. Στην πολιτική για το γάλα έχουμε πλεονάσματα και λόγω των, ε, της μείωσης των ποσοστώσεων. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει πάλι η αγορά του γάλακτος. Μήπως πρέπει να εισάγου, εισαγάγουμε πάλι κανόνες ε, για την ε, αγορά. Ε, τρεις ερωτήσεις συγκεκριμένες τώρα. Καταρχήν τα εσπεριδοειδή στη Βαλένθια. Και... ρόδια και αν ε, ε, μπορούν να υποστηριχθούν αυτά τα προϊόντα μετά τα προβλήματα. Επίσης τα 4 ε, εκατομμύρια για την κρίση επαρκούν και πώς θα επιδράσουν στις άμεσες ενισχύσεις και πώς θα επηρεαστούν μάλλον οι άμεσες ενισχύσεις μετά από αυτούς τους παραγωγούς. Επίσης το εμπόριο τώρα ακόμα και με την κρίση κερδίζει οι τιμέ για το βουτυρό στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 20% από μεγάλες αλυσίδες ε, εμπορικών καταστημάτων. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό με τις μεγάλες αλυσίδες ούτως ώστε να μην αυξάνεται το κέρδος ε, των εμπόρων σε περίοδους κρίσης. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει παρόμοια προβλήματα, πρέπει όμως να είμαστε πολύ ρεαλιστές στη σημερινή μας συζήτηση. Πρόκειται για την ε, απαρχή ε, μιας μεγάλης διαμάχης ε, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ε, θα δούμε περικοπές στις τιμές, αλλά δεν θα πρέπει να συμβάλλουμε και να ενθαρρύνουμε την ε, ε, απεσιοδοξία στην αγορά. Θα πρέπει να λάβουμε θετικά μέτρα. Ένα θετικό μέτρο ε, είναι ένα ζήτημα είναι η, εξαφάν, η κατάργηση των ποσοστώσεων. θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά. ορισμένα κράτη-μέλη προετοιμάζουν την αντίδρασή τους και αυξάνουν την παραγωγή. Οι τιμές παρέμβασης τώρα ε, είναι τελείως μη ρεαλιστικές και δεν αντιπροσωπεύουν αυτά που χρειάζεται η αγορά. Τι θα κάνει η Κομισιόν, θα αυξήσει την τιμή παρέμβασης και θα δείξει καλή θέληση σε αυτό το τομέα, αν χρειαστεί. Πέρσι είχαμε τη δέσμη των γαλακτοκομικών. Ε, τώρα υπάρχουν τα εργαλεία στη διάθεσή σας για να γίνει η δουλειά που πρέπει και που είναι τόσο σοβαρή τους επόμενους μήνες. Τέλος, ε, εντάξει με την ιδιωτική αποθεματοποίηση, όμως ε, αν πάνε προϊόντα στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, τον επόμενο Μάρτιο όταν θα ε, αρχίσει η παραγωγή ε, πώς θα απολυθούν δηλαδή θα ληφθούν υπόψη, ε, θα δοθούν μεγαλύτερα ε, χρονικά διαστήματα ε, κατά τα οποία τα προϊόντα θα έχουν μπει στην ιδιωτική αποθεματοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Μπιτσότο υπόθηκε ότι η απαγόρευση χτύπησε με διάφορους τρόπους τα κράτη-μέλη, αλλά υπόθηκε ότι το ίδιο ισχύει και για διάφορες περιφέρειες εντό των κρατών. Στην περιοχή του Βένετο μέχρι τώρα η ζημιά είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά. Είναι γελία τα ποσά που έχουν ε, τεθεί στη διάθεση για αποζημιώσεις. Έτσι λοιπόν ζητώ από τους συναδελφούς να υπάρχει ουσιαστική δέσμευση, όχι όπως έγινε μέχρι τώρα. Επίσης σας ζητώ να Είμαστε αποφασισμένοι και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει αυτές τις κυρώσεις γιατί δεν μπορούν οι Γεωργοί να πληρώνουν τις λάθος επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν συνεχίσουμε έτσι η κρίση θα γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη το να ε, αυξάνουμε τις κυρώσεις ε, είναι πραγματική τρέλα και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να την πληρώσουν οι Γεωργοί. bardzo, panie przewodniczący. Ja także chcę zwrócić uwagę. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω, λέει ο κύριος Κουτσμιούκ, ότι όταν πρόκειται για την υποστήριξη των ε, παραγωγών οποροκυπευτικών, θα πρέπει να φτάσει στους ε, μεμονωμένους παραγωγούς η βοήθεια, αυτούς που και να βοηθήσουν αυτούς που είτε διαθέτουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς τα προϊόντα είτε τα δίνουν για να καταστραφούν. Θα πρέπει να υποστηριχθεί το εισόδημά τους λόγω επίσης των μεγάλων ε, μειώσεων των τιμών. Θα πρέπει η Κομισιόν υποβάλει ένα πρόγραμμα στήριξης για αυτούς που έχασαν τα εισοδήματά τους. Χωρίς τη λύση αυτή η υποστήριξη θα είναι συμβολική μόνο. Και ένα δεύτερο θέμα είναι η κατάργηση των ποινών για την υπέρβαση των ποσοστώσεων. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η αγορά τώρα που οι πρόσθετες αυτές κυρώσεις είναι απόλυτα κατανόητες. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ ναι. κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς πολύ κύριε Κόρτε που διαφωτίσατε την Επιτροπή μας. Όμως με λίγο που ο Επίτροπος Γεωργίας δεν είναι παρόν ε, ίσως ε, έχει κάποια άλλη υποχρέωση ή ασθενή ή δεν ε, ενδιαφέρεται πια να συνεργάζεται μαζί μας. Πάντως θα πρέπει να κάνουμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που ε, λάβατε. Αυτά συμπεριλαμβάνουν και καλά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρξει ταχεία δράση για τα ευπαθή προϊόντα καταρχήν και για τα αποβουτυρωμένο, το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη και εκεί χρειάζεται γρήγορη ε, παρέμβαση για να αποσυμφορηθεί η αγορά. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε τα ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα τα οποία τώρα ε, ε, δεν εξάγονται στη Ρωσία να ε, με ειδικές διαδικασίες να ε, εξαχθούν σε άλλες χώρες. Θα πρέπει όμως να αναλυφθεί άμεση δράση για να αποσυμφορηθεί όπως σας είπα η αγορά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βοητσοκόφσκι. Θέλω να ρωτήσω γιατί η Κομισιόν δεν χρησιμοποίησε κονδύλια από το Ταμείο για τις κρίσεις, ε, γιατί εκτός από αυτά τα 400 εκατομμύρια ε, αυτά έχουμε αυτά ε, προέρχονται από τις, ε, τους κανονισμούς για την κοινή οργάνωση της αγοράς για να αντιμετωπιστούν τις λειτουργίες στην αγορά. Υπάρχουν τις λειτουργίες στην αγορά. Σε άλλες χώρες Είχαμε σοβαρή κρίση όμως όπως στις βαλτικές δημοκρατίες, τη Φιλανδία, την Πολωνία, ως ένα βαθμό τη Γερμανία. Αυτές είναι οι χώρες που επλήγησαν ως επιτοπλίστων από το εμπάργκο και τώρα ε, μπήκαν σε σοβαρή κρίση. Άρα πρέπει από το Ταμείο για τις Κρίσεις να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια και τώρα πηγαίνουν στα κράτη-μέλη. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί όταν έχουμε βακτήρια ε κόλλη ε, μπορούσε, μπορούσε η, Κομισιόν να αντιδράσει γρήγορα και να, δώσει, να κάνει τις πληρώμες. Τώρα έχουμε μια σοβαρότατη γεωργική κρίση ε, τους πρόσφατους πρόσφατου, τώρα και δεν βάζετε χέρι σε αυτά τα κεφάλαια, δεν τα χρησιμοποιείτε, δεν τα διαθέτετε. Ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όμως γιατί η κρίση είναι σοβαρότατη. Η κυρία Χράνς Καρσία. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι αυτή την περίπτωση έλαβε δράση πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν και αυτά τα 125 εκατομμύρια ευρώ φαίνονται καλά για αρχή. Νομίζω ότι θα έπρεπε όμως να είχαμε υπάρχει οικονομική διαθεσιμότητα για τις μελλοντικέ ανάγκες που θα έρθουν ε, με ε, την ε, παραγωγή εσπεριδοειδών και άλλων προϊόντων. Επίσης, θέλω να πει η Κομισιόν έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα ντόμινου, παραδείγματο χάρη η Πολωνία εξάγει μανιτάρια ε, στην ε, Ρωσία. Όταν ε, όμως θα πλημμυρίσει αυτό το μανιτάρι της ευρωπαϊκής αγοράς, τι θα γίνει. Επίσης, νέες αγορές, τι μπορούμε να κάνουμε, παραδείγματο χάρη, για να φτάσουμε στην Αμερικανική αγορά, να μας εμποδίζουν τα φυτογειονομικά μέτρα. Επίσης, η Πολωνία πρότεινε να πάμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το λαμβάνει σοβαρά αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια μέτρα σκέφτεται να λάβει εν ώψη του ΠΟΕ. Η κυρία Αγγιλέρα, ευχαριστώ. Συζητάμε τις συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Γεωργία που προήλθαν από τι πολιτικέ αποφάσει που θετήθηκαν κατευθείαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πρόκειται για μια πολιτική διένεξη που όλοι ελπίζουμε να λήξει σύντομα, όμως οι προοπτικές ε, δεν είναι και τόσο αισιόδοξε, γι' αυτό όλα αυτά μας ανησυχούν. Η Κομισιόν μας ζητά να υποστηρίξουμε τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί. Κατά την άποψή μου, για να τα υποστηρίξουμε θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά δίκαια και ισορροπημένα. Αποτελεσματικά αν είναι χρήσιμα για τον κλάδο. Χρήσιμα δηλαδή να λύνουν τα προβλήματα για όλο το γεωργικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να προβλέπουν μηχανισμούς ε, πρόβλεψης κρίσεων ώστε να μην πέφτουν τιμές. Επίσης, ε, πρέπει να έχουμε και ημερομηνία λήξης. Όταν θα λήξει το βέτο, θα πρέπει να λήξουν και τα μέτρα και θα πρέπει να είναι δίκαια. Και να πω για τη δική μου χώρα και για περιφέρειες της δική μου χώρας όπως η Μούρση, η Ενδελουσία, η Βαλένσια, η Καταλωνία, η Αραγωνία, η Καστίγια Λεόν, η Καστίγια Λαμάντσα, Έχουμε πολύ μεγάλη επιδείνωση της κατάστασης. Έχουμε πολύ μεγάλη... πολύ μεγάλο πρόβλημα σε κάποιες υπηρετικές καλλιέργειες ε, βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για αυτές τις καλλιέργειες, αλλά δεν ε, υπάρχει ευαισθησία απέναντι στα σπεριδοειδή, το χάρη, γιατί το χάρη δεν λαμβάνεται υπόψη τις περιπτώσεις του καρπουζιού, του πεπονιού κτλ. Παρακαλώ πρόεδρε, έχω ακόμη χρόνο και ε, για τα λαχανικά. Γιατί το χάρη βάζετε το αγκούρι και τη μελιτζάνα, όχι, δεν καταλαβαίνω ποια είναι τα κριτήρια, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία λοιπόν όλα όσα δεν πάνε στη ρωσική αγορά δημιουργεί κάποιες συνέπειες και στις λοιπές παραγωγές. Δηλαδή εδώ πρέπει να έχουμε και μία εκστρατεία προώθησης για την εσωτερική κατανάλωση. Πρέπει να το κάνει αυτό η Κομισιόν και πρέπει η Κομισιόν να αναλύσει τι γίνεται με, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ε, τελικά εποφελείται από αυτή την κρίση και ζημιώνονται περισσότερο οι Ευρωπαίοι γεωργοί. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Ο Σταραμπέλα, Ταραμπέλα, ευχαριστώ. Το περασμένο Σαββατό ε, είχα πάει στη Λαϊκή και εκεί εγώ ήθελα να προωθήσω την τοπική παραγωγή και έκανα τον πολιτή μήλων και τελικά ενημερώθηκα τι συμβαίνει με τον κίνδυνο της καταστροφής. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλο Σε Αυτός πρέπει να το αποφύγουμε. Εμείς δεν θα έπρεπε να υποφελούμαστε από αυτό το εμπάργκο της Ρωσίας και να το δούμε μια ευκαιρία για να επιμείνουμε στην αναγκαιότητα ε, για τα προκυπευτικά να καταναλώνουμε περισσότερο και να δώσουμε μια νέα όθηση στην εσωτερική αγορά. Γιατί ξέρετε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία λέει ότι τουλάχιστον πρέπει να τρώμε 400 γραμμάρια φρούτα την ημέρα και υπάρχουν πολύ λίγε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πετύχει αυτό το στόχο. Έτσι λοιπόν, εγώ το βλέπω αυτή την ευκαιρία ότι μπορούμε να κάνουμε μια εκστρατεία ε, για να καταναλώνουμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά που είναι πολύ καλά για τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ κύριος Καλινόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, είπατε ότι το πλήγμα είναι πολύ σοβαρό. Αν όμως δούμε τα ποσά που χρησιμοποιούνται στην παρέμβαση και αν τα συγκρίνουμε με τα ποσά που διατέθηκαν στην κρίση του ε κόλλη, βλέπουμε, αποκομίζουμε την εντύπωση ότι το θέμα δεν το βλέπει τόσο σοβαρά η Κομισιόν, ενώ είναι τόσο σοβαρό γιατί είναι χιλιάδες οι αγρότες που είναι σε κακή κατάσταση. Προκειμένου περί του γάλατος συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι πρέπει να καταργήσουμε κάποιες ε, κυρώσεις για αυτούς που υπερέβησαν τις ποσοστώσεις. Αλλά μην κάνουμε διακρίσεις μεταξύ αυτών που ανήκουν σε οργανώσεις παραγωγών και των άλλων. Δεν μπορούμε να τιμωρούμε τους ε, ανεξάρτητους παραγωγούς. Αναφέρατε κάποια προϊόντα που δεν θα συνεπάγονται κυρώσεις, ε, λάχανο κλπ. Ε, υπάρχουν πολλές κατηγορίες όμως ε, λάχανων. Ε, είναι πολλά τα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν στον κατάλογο των αποζημιώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur le Président. Euh, en tant que député, mais aussi en tant que γεωργός και βουλευτής, γιατί παράγω λαχανικά, γνωρίζω λίγο τα πράγματα και πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Με βάση αυτά που μας είπε η Κομισιόν έχω μερικά ερωτήματα. Πρώτον, χαιρετίζω την τη γρήγορη αντίδραση του Επιτρόπου Τσόλος, αλλά είναι ανεπαρκή τα μέτρα. Σίγουρα θα ληφθούν και συμπληρωματικά αλλά όπως αναρωτιέται και η ίδια η Κομισιόν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με ορισμένα φραγμούς όπως την τιμή απόσυρσης που χρησιμοποιείται με τρόπο τελείως ανισομερή. Ορισμένα προϊόντα δεν έχουν αποσυρθεί καθόλου γιατί η τιμή απόσυρσης είναι πολύ πολύ μακριά από το κόστος παραγωγής το ίδιο. Άλλο θέμα, επίσης τεχνικό, το μέτρο de minimis. Τέλος, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, αλλά να ζητήσουμε από τους γεωργούς να συγχρηματοδοτήσουν τέτοια προώθηση κατανάλωσης είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε. Thank you. Thank you, Chairman. Uh, I regret that... Uh, Ευχαριστώ. Ε, δυστυχώς ε, δεν υπάρχει διερμηνία στα φιλανδικά, ενώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για τους φιλανδούς ε, γεωργούς και τη γεωργία μας. Τέλος πάντων, ε, ήταν αναπόφευκτη η ανακλιμάκωση των κυρώσεων μετά την ε, στάση της Ρωσίας στην Ουκρανική κρίση. Ε, όμως ε, η επίδραση της απαγόρευσης είναι διαφορετική στις χώρες μέλη. Υπάρχουν ορισμένοι, όπως οι χώρες της Βαλτικής, η Φιλανδία, η Πολωνία, εκεί οι απώλειες είναι πολύ σημαντικές. Είναι σημαντικό λοιπόν να, να φροντίσει ε, και να αντιμετωπίσει η Κομισιόν τις δυσκολίες ε, των γεωργών, γαλακτοπαραγωγών με αποτελεσματικά μέτρα καλύπτοντας, ε, ε, ε, χρησιμοποιώντας όλο το οπλοστάσιο που διαθέτει όπως αναφέρθηκε και υπογραμμίστηκε άλλωστε. Θα πρέπει να ελαφρύνει το πρόβλημα των παραγωγών ούτως ώστε οι απώλειες να μην γίνουν υπερβολικές δυσβάστακτες και η Ένωση θα πρέπει να φροντίσει αυτούς που επλήγησαν ως επιτοπλίστων από την απαγόρευση των εισαγωγών θα πρέπει να είναι επαρκής η υποστήριξη και χρειάζεται ταχεία ανάληψη δράσης. Αυτή η αλληλεγγύη είναι σημαντικό ε, να υπάρχει, ούτω ώστε να υπάρχει και δημόσια στήριξη της γενικότερης πολιτικής μας ανάσχεσης. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να είναι σήμερα παρόν ο Επίτροπος, δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση κανονικά, ο Επίτροπος πρέπει να φροντίσει να μας συναντήσει. Οι επιπτώσεις ε, ε, μας επηρεάζουν και στην δική μας την περίπτωση. Ε, η, κοινή η κινήμη της ντομάτας στην περιοχή μου έχει πέσει πάρα πολύ. Επηρεάζονται λοιπόν πολλοί τομείς της αγοράς. Ε, πρέπει να ε, προβλέψουμε για το γεγονός ότι δεν θα επαρκέσουν τα κονδύλια. Ε, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό. Και τέλος θα έπρεπε να απευθύνουμε επιστολή στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ούτως ώστε να πιέσουν για την αύξηση των δημοσιονομικών κονδυλίων. Ρώτηση στην Κομισιόν για τα προγράμματα για τα σχολεία. Το είπα και χθε. αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να προβληθούν για να αξιοποιηθούν, να μειωθεί και η γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ε, επίσης, ε, η σταθεροποίηση του εισοδήματος είναι πολύ ε, σημαντική για μεγάλη μερίδα των γεωργών. Ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τα λάθη του παρελθόντος ε, όταν ε, ε, κάναμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και τότε όλοι θέλαμε να καταργήσουμε όλες τις παρεμβάσεις. Εμείς σήμερα ζητάμε νέες παρεμβάσεις από την Κομισιόν. Το πακέτο κατά της κρίσης που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθύμησε ο κύριος Δεντέν και άλλα. Εμείς ε, το οικοδομήσαμε χωρίς ε, πόροι και σήμερα οι γεωργοί θα πληρώσουν τις συνέπειες, ε, δηλαδή το γεγονό ότι δεν υπάρχουν πόροι και τελικά η δημοσιονομική πειθαρχία θα μας οδηγήσει στο να πληρώσουν οι γεωργοί. Τώρα, είπατε για το τυρί έχουμε 33% του τυριού να εξάγεται στη ρωσική αγορά. Μιλάμε για τεράστια αγορά. Με την ιδιωτική θεματοποίηση ρισκάρουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα μεταξύ των τυριών που έχουν ονομασία προέλευσης ε, σε σχέση με άλλα. Έτσι λοιπόν θέλω να εξετάσει η Κομισιόν αυτό τον ε, κίνδυνο στρέβλωσης μπορεί να υπάρχει γιατί αυτά τα είδη των τυριών δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ο Η Κομισιόν μας τόνισε ότι τα τρόφιμα που πουλούσαμε στη Ρωσία πρέπει να πουληθούν κάπου αλλού και οι πολίτες της Ρωσίας που δεν θα έχουν αυτά τα τρόφιμα και αυτοί επίσης πρέπει να βρουν τρόφιμα από αλλού. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι οι μεσάζοντες εποφελούνται. Ζητώ από την Κομισιόν να μην μειώσει αυτό το καινούριο εμπόριο που θα δημιουργηθεί μέσω της γραφειοκρατικής διαδικασίας που θα επιβάλλει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω τις επιπτώσεις που θα έχουν οι κυρώσεις για τη Ρωσία στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων στην Ένωση. Και επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για τις αποζημιώσεις που πρέπει να δώσουμε και να υπολογίσουμε πώς θα, πού, πού θα τις βρούμε και πού θα τις διαθέσουμε. Όχι απλοϊκά, μόνο με τον όγκο δηλαδή προϊόντων που θα απολούνταν στη Ρωσία, γιατί θα μπορούσαμε να ζημιωθούμε και αν ορισμένες παραγγελίες ακυρωθούν στην κοινοτική αγορά μέσα στην Ένωση γιατί όλα τα προϊόντα που θα παραμείνουν στο εσωτερικό της Ένωσης θα στρεβλώσουν την αγορά. Παραδείγματο χάρη η Ρουμάνη παραγωγή που πουλούσαν τα προϊόντα τους στη Γερμανία θα διαπιστώσουν ότι η γερμανική αγορά θα είναι υπερπλήρης φέτος και θα υπάρξουν τεράστια αποθέματα για τη Ρουμανία. Οι παραγωγοί μας έχασαν περίπου τη μισή τους σοδιά. Άλλες χώρες που έχουν ζημιωθεί επίσης από τη ρωσική αγορά, εμείς χάσαμε από την ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη, όχι μόνο τις πωλήσει προς τη Ρωσία και γι' αυτό ζητώ να το σκεφτεί και αυτό η Κομισιόν. Ο κύριος Δενόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω μια μαρτυρία. Είμαι πρόεδρος της περιφέρειας του Λιμουζέν στη Γαλλία που είναι γεωργική περιφέρεια και είχε πολλές εμπορικές σχέσεις με δύο ρωσικές περιφέρειες για τα γεωργικά προϊόντα συγκεκριμένα και διαπίστωσα πηγαίνοντας επιτόπου στη Ρωσία πολλές φορές ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση της Ρωσίας και των Ρώσων για γεωργικά προϊόντα από τη Γαλλία αλλά και από άλλες χώρες της Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν αυτές οι κυρώσεις γιατί θα βλάψουν και τον λαό της Ρωσίας και την Ένωση. Στην περιφέρειά μου διαπιστώνω ότι χίλιες αγελάδες που θα εξάγονταν στη Ρωσία η παραγγελία έχει ακυρωθεί και αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στους παραγωγούς. Πρέπει η Κομισιόν δηλαδή να αρχίσει να το σκέφτεται και αυτό και την αγορά κρέατος αλλά και λαχανικών. Η Ρωσία τα χρειάζεται και επομένως δεν θα κρατήσει και πολύ το μέτρο. Και για το γάλα τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Κάμπ Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για μια μεγάλη παγκόσμια κρίση. Κλιματική, ε, βιοκαυσίμων, καυσίμων, ε, τροφίμων ότι θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που έχει ο πλανήτης, ο οποίος φλέγεται και θα πρέπει γι' αυτό να ληφθούν ε, νυφάλιες αποφάσεις ε, με βάση τα διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος. Το παράδειγμα εν προκειμένου του κυρίου Ταραμπέλα είναι πάρα πολύ θετικό θα πρέπει να βρούμε καινούριου δρόμους πρόθεσης των απορροκυπευτικών. Δεν ξέρω, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αύξηση της παραγωγής σε μια δύσκολη περίοδο όπου ήδη οι δυνατότητες του πλανήτη έχουν αρχίσει να εξαντλούνται, ε, θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, δηλαδή μικρές αποστάσεις, ε, και υποστήριξη των γεωργών για την βιώσιμη παραγωγή. Όπως σας είπα, των σύντομων διαδρομών, αποστάσεων. Ενδεχομένως ε, τα βιολογικά προϊόντα θα έπρεπε να διατίθενται και σε αγορές των τρίτων χωρών ή θα υπάρξουν αρνητικές ε, επιπτώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι και εγώ για την απουσία του Επιτρόπου σήμερα. Ε, σι... Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν παρόν και στην ΚΟΠΑ ήταν παρόν. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, είχε παρουσιάσει τα μέτρα. Ε, η Ολλανδία φύγεται, πλήττεται πάρα πολύ. Τα 125 εκατομμύρια ε, μάθαμε από το καλοκαίρι ότι θα ήταν διαθέσιμα, αλλά δεν φτάνουν, χρειάζονται περισσότερα κονδύλια και θα δοθεί ένα μήνυμα μέσα από τον προϋπολογισμό για όλους τους τομείς και για το χείριο κρέας, αφού όλοι οι τομείς στην Ευρώπη πλήττονται. Και συμφωνώ πάνω σε αυτό με τους προηγούμενους ε, συναδέλφους. Και τα προγράμματα στα σχολεία είναι σημαντικά ε, ελπίζω ότι γρήγορα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη, τη, με τα μέτρα μας τη, το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Σφερά. Να δύο παρατηρήσεις, ε, ουσιαστικές αλλά από ε, το τύπο. Να έχουμε την πιο σοβαρή πολιτική κρίση από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να λάβουν κάποια αντίπεινα κατά της Ρωσίας. Εγώ Νομίζω ότι το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να περάσει από μια ανάπτυξη πολιτική στρατηγική ισχυρή με τη Ρωσία. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρώπη ε, θα κοστίσουν ακριβά και έχω την εντύπωση εδώ ότι είμαστε κάπως σαν πυρομανείς πυροσβέστες. Η Γαλλία ε, σήμερα ε, ε, ουσιαστικά χάνουμε όλα αυτά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Τελικά, αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, εγώ πρέπει να σκεφτώ τους Γάλλους γεωργού αλλά και του Ευρωπαϊού γεωργού και νομίζω ότι δεν έχει δράσει υπεύθυνα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κρίση και ε, δεν μπορεί να αναλάβει τις συνέπειες ε, μιας επιλογής που ξεκίνησε εδώ και κάποιου μήνε. Παρακαλώ. κύριε Μαγκίνες. Εγώ υποστηρίζω αυτούς που καλούν την ανάληψη δράσης για το γαλακτοκομικό τομέα. Τώρα είμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, εξετάσει εκ νέου το Συμβούλιο το θέμα της υπερισφοράς. Εγώ νομίζω ότι οι κύριοι Νταντέν και Ντεκάστρου έκαναν κάποιες πολύ κατάλληλες παρατηρήσεις σήμερα το πρωί. Θέλουμε περισσότερα από αλληλεγγύη μεταξύ των γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε αλληλεγγύη για τους γεωργούς στην κρίση ναι. αυτή από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αγροτική η κρίση αυτή, είναι πολιτικό πρόβλημα και επομένως πρέπει να πιέσουμε στην Επιτροπή μας για επαρκείς πόρους και αυτό σημαίνει πέρα, πόρους πέρα από όσους υπάρχουν σήμερα στον προπολογισμό για τη γεωργία προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην αγορά. Το τρίτο σημείο το ανέφερε ο κύριος Μέλο, πρόταση να μειώσουμε άμεσα τις πληρωμές ε, στους γεωργούς για να δώσουμε αποζημίωση σε κάποιους άλλους γεωργούς είναι απαράδεκτη. Γιατί ήδη έχουμε περιορισμένο προϋπολογισμό για τις άμεσες πληρωμές και τις άμεσες ενισχύσεις ε, και εγώ νομίζω ότι πρέπει η Κομισιόν να τοποθετηθεί στο έτοιμά μας για περισσότερους πόρους. Ευχαριστώ, Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί και εγώ ήθελα να πω αυτό που μόλις τώρα είπε η κυρία Μαγκίνες. Αυτή η κρίση δεν προέρχεται από τη γεωργία, είναι μεγάλη διεθνής κρίση και τις συνέπειες τις πληρώνει η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ε, αυτό δεν το επιλέξαμε εμείς, έτσι αποφάσισε η Ρωσία. Στα πλαίσια του γεωργικού προϋπολογισμού αναζητούμε τώρα πόρους που δεν επαρκούν και εν μέρη δίνουν γελία αποτελέσματα όπως η τιμή της παρέμβασης που δεν καλύπτει ε, τα, τα, τα προϊόντα και την παραγωγή τους και γενικά η αγορά της παρέμβασης δεν δίνει λύση. Πρέπει λοιπόν να επιδείξουν όλοι αλληλεγγύη και θα πρέπει και το Σώμα των Επιτρόπων και ο Επίτροπος Γεωργίας να βρουν άλλα ε, κονδύλια, όχι μόνο μέσα από τον ε, γεωργικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ κυρία Μόη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν γνωρίζει ε, το εξής. Ε, το ότι οι γεωργοί πραγματικά έχουν γονατίσει κυρίως στην Νότια Ευρώπη, γιατί χωρίς κανένας έλεγχος ποιότητας σε πολύ χαμηλές τιμές έρχονται τώρα και μας κατακλείζουν τα προϊόντα από το Μαρόκο. Επίσης ε, έχουν φτάσει οι γεωργοί σε σημείο να μην θέλουν ε, καν ε, να συλλέξουν τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν πέρα από το θέμα της Ρωσίας υπάρχει και αυτή η κατάσταση που σας ανέφερα που ισχύει εδώ και καιρό. Υπάρχει κάποιο σχέδιο από την Κομισιόν για να βοηθήσει αυτούς τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά συμμερίζομαι όσα υπόθηκαν. Η κρίση αυτή είναι κυρίως πολιτική. Η Κομισιόν έχει καταφέρει πάντως και τη συγχαίρω γι' αυτό να παρέμβει γρήγορα από τον Αύγουστο ήδη. Είναι πολιτική και υπόθηκε επίσης ότι την ύφη την πληρώνει η Γεωργία και η Γεωργή. Το θέμα που τίθεται εδώ είναι η διαχείριση βραχυπρόθεσμα αλλά και η πρόβλεψη του προσωπρόθεσμου. Το βασικό πρόβλημα, το είπαν και άλλοι αλλά το υπενθυμίζω και εγώ, είναι τα μέσα και τα κονδύλια. Η κρίση αυτή μας υποχρεώνει να θέσουμε το θέμα ειδικών προϋπολογισμών για αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Αυτό λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και μεταξύ μας. Αλλά σε τι χρονοδιάγραμμα, τι προβλέπει η Κομισιόν, πότε προβλέπει η Κομισιόν να μπορέσει να γίνει μια τέτοια συζήτηση, γιατί μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ρίξον. Ευχαριστώ. Να πω μόνο ότι πιστεύω ότι η Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα, σωστά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο για κάποιες περιφέρειες, για κάποιους γεωργούς στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι υπερβολικό να μιλάμε για κρίση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Πολλοί υπερτονίζουν τη διάσταση της κρίσης. Δεν είναι τόσο πολύ πιστεύω. Φυσικά πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη με τους πληγέντες, αλλά μακροπρόθεσμα και στην παγκόσμια αγορά δεν νομίζω ότι θα ε, υπάρξει πτώση των τιμών και νομίζω ότι πολλά προϊόντα θα μπορέσουν να απολυθούν αλλού, σε εναλλακτικές αγορές από τις τωρινές. Ευχαριστώ, Ριμπέλο. Ανησυχώ πάρα πολύ με τα αποτελέσματα του ρωσικού εμπάρου όχι μόνο για τα άμεσα αλλά και τα άμεσα αποτελέσματα θα πρέπει να αποφύγουμε μια χιονοστιβάδα που θα πλήττει όχι μόνο τα κρατημέλη που εξάγουν περισσότερο στη ρησία αλλά και όσοι θα υποφέρουν ε, από ε, τις απαντήσεις που θα δοθούν ε, από άλλους η απάντηση ευρωπαϊκή πρέπει να αξιολογηθεί αλλά και δική μας ικανότητα να ε, προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα ιστορικά μας προβλήματα και αυτό που είχαμε όπως με το γαλακτοκομικό τομέα ποια μέτρα θα πλάβει η Κομισιόν για τα κρατημέλη που έμεσα θα πληγούν όπως η Πορτογαλία που δεν έχουν οικονομική ικανότητα για να δώσουν μία απάντηση μέσω κρατικών ενισχύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 35 ομιλητές παρενέβησαν στη συζήτηση αυτή. Και τώρα κύριε Κόρτε έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να παραδεχτώ ότι δεν θα μπορέσω να απαντήσω στα πάντα. Αυτό που έκανα με τη βοήθεια των συναδέλφων είναι να ομαδοποιήσω ε, τις ερωτήσεις σε πέντε ομάδες. Οπότε να προσπαθήσω να καλύψω ε, τις ερωτήσεις από τις ομάδες. Το πρώτο μήνυμα που πήρα καθαρά από πολλά αξιότιμα μέλη είναι ότι δεν κάναμε αρκετά. Αυτό προέκυψε ως αφέστατο αποτέλεσμα. Τι να πω πάνω σε αυτό. Πρώτον, αλήθεια είναι ότι ε, το πλωστάσιο για την κρίση που το, έτσι το είπα και έτσι το είπε και ο Επίτροπος, ε, καλύπτουν ε, ε, όλα αυτά ε, τώρα πρόκειται να δοκιμαστούν για πρώτη φορά το δίχτυ ασφαλείας κλπ. Η προσέγγιση του Επιτρόπου Τσιόλος είναι ότι πρέπει να τα δοκιμάσουμε όλα αυτά και είπε αν αυτά δεν είναι αρκετά θα κάνουμε περισσότερα. Ας χρησιμοποιήσουμε καταρχήν λοιπόν τα υπάρχοντα εργαλεία μας, τους μηχανισμούς μας και αν δεν επαρκέσουν εδώ είμαστε για να κάνουμε περισσότερα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στις αγορές και θα αντιδράσουμε όταν υπάρξει ανάγκη. Και έτσι περνάω στον κατάλογο για τα αγροτυπευτικά για παράδειγμα που δεν είναι, ε, ισορροπημένος, είπαν ορισμένα αξιότιμα μέλη. Γνωρίζουμε βέβαια ότι τα εσπεριδοειδή ή άλλα προϊόντα από τη Νότια Ευρώπη δεν είναι στον κατάλογο. Δεν μπήκαν στον κατάλογο γιατί η συγκομιδή θα λάβει χώρα αργότερα μέσα στον χρόνο αλλά δεν είπαμε ότι δεν θα κάνουμε κάτι για αυτά τα προϊόντα. Τα μέτρα που πήραμε στα μέσα Αυγούστου θα καλύψουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για 125 εκατομμύρια ευρώ και θα δούμε πολύ προσεκτικά τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα. Και αν χρειαστεί να λάβουμε μέτρα για τα λάχανα, τα εσπεριδοειδή και κάποια άλλα προϊόντα που αναφέρθηκαν, βεβαίω και θα λάβουμε για να τα καλύψουμε. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, για αυτό που είπε για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, το ύψος της ενίσχυσης και τη διάρκεια. Ο κύριος Νίκολς το είπε. Η διάρκεια ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τα τυριά, όχι μόνο, όχι, και για το βούτυρο και για το αποκορυφωμένο γάλα, είναι αυτή που πάντα χρησιμοποιούσαμε. Ε, ανέκαθεν αυτά τα ποσά χρησιμοποιούσαμε και στηρίζονταν στο κόστος αποθεματοποίησης, ε, τα στοιχεία που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη, που είναι αξιόπιστα. Θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αν δούμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Θα το δοκιμάσουμε. Η 7 μήνη περίοδος που αναφέρατε και που είναι σωστή μπορεί να παραταθεί πρώτον, αλλά πρέπει να εξηγήσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα τυριά ή μάλλον τα τυριά που μπήκαν στην ε, αποθεματοποίηση την ιδιωτική το Μάρτιο θα εξακολουθούν να ε, εποφελούνται. Είναι 7 μήνες. Δηλαδή δεν είναι αυτά που είναι τώρα στην αγορά, μόνο αυτά τα εταιριά θα ωφεληθούν. Το πρόγραμμα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι θα νόμιζε κανείς πάνω στη βάση του κανονισμού. Δεύτερον, ε, ο προϋπολογισμός. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά τα μέτρα. Και δεν πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό και μήπως χρειάζεται το αποθεματικό ή το Ταμείο για τις Κρίσεις. Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα, πολύ δύσκολο και νιώθω κάποια αμηχανία και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες πρώτον γιατί το τοπίο είναι ασαφές. Μπορώ να πω ότι οι τωρινές, οι τρέχουσες δαπάνες που έχουμε αναλάβει, τα μέτρα που έχουν καταγραφεί, χρηματοδοτούνται όλα από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό. Δεν έχουμε αποφασίσει δηλαδή να ανοίξουμε τη διαδικασία ε, χρησιμοποίησης του Ταμείου για τις κρίσεις. Μπορεί να γίνει αυτό αργότερα. Όχι ε, μέσα στον προϋπολογισμό του 2014 που ε, στην ΚΑΠ ολοκληρώνεται, τελειώνει στις 16 Οκτωβρίου για τον απλό ρόλο ότι δεν αναμένουμε οι αδίποτε από αυτές τις δαπάνες που γίνονται να δηλωθούν σε μας πριν από την ημερομηνία αυτή. Οπότε θα έχουμε τα πρώτα τιμολόγια των κρατών μελών μετά τις 16 Οκτωβρίου. Και αυτό σημαίνει ότι εμπίπτουν πια στον προϋπολογισμό του 2015. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα προϋπολογισμός του 2015. Το μόνο που υπάρχει τώρα είναι μια πρόταση από την Κομισιόν που νομίζω ότι είναι για 58 εκατομμύρια ευρώ για την ΚΑΠ. Όλα τα μέτρα μαζί. 58 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πρόταση. Αλλά εσείς και το Συμβούλιο είσαστε η αρχή επί του προϋπολογισμού και οι αποφάσεις ε, τροποντινά ως ένα βαθμό είναι δική σας. Μέχρι να ξέρουμε πόσα χρήματα θα υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 2015 ε, πριν από αυτό δεν μπορούμε να ε, μιλάμε για το Ταμείο για τις Κρίσεις. Νομίζω ότι και πολιτικά είναι πιο πιστικό επιχείρημα να αρχίσουμε όταν έχουμε τον το ποσό για τον προϋπολογισμό του 2015 και μετά θα δούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει επί τόπου, δεν, ξέρω τι... Ε, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Αυτά μόνο έχω να πω τώρα ε, πάνω σε αυτό. Και κάτι ακόμα. Κάποιο αξιότιμο μέλος είπε ότι ε, μόνο οι αγρότες πλήττονται από τις κυρώσεις. Αυτό ισχύει στο βαθμό που μιλάμε για το άμεσο εμπάργο, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας που πλήττονται από την κρίση αυτή. Και αν διαβάσετε τις εφημερίδες θα δείτε ότι δεν πρόκειται μόνο για τους αγρότες. Ε, γαλακτοκομικά πολλά, είπατε για αυτά, χαμηλές τιμές παρέμβασης, παραμονή της ποσόστοσης, θα πρέπει να γίνει, ε, γίνουν διορθώσεις και εδώ ε, θα πω πάλι το ίδιο ότι πρώτα θέλουμε να δούμε και να δοκιμάσουμε τα συστήματα που υπάρχουν. Ε, από νομοθετικά έχουν θεσπιστεί οι τιμές παρέμβασης σε ένα χαμηλό επίπεδο, αλλά αυτό επειδή οι τιμές ήταν επί σειρά ετών πολύ υψηλέ. Ήταν πολύ ανθυρή, ανθυρός ο γαλακτοκομικός τομέας για αρκετά χρόνια. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά μέσα σε μια προοπτική. Αλλά και πάλι δεν αποκλείουμε τίποτε. Οι ποσοστώσεις ε, θα καταργηθούν του χρόνου το Μάρτιο, η απόφαση αυτή πάλι έχει ε, ληφθεί νομοθετικά. Ε, για τις διορθώσεις ε, είχαμε δύο-τρεις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή πολιτική υποστήριξη ούτως ώστε να αλλάξει το ποσό της διορθώσης. Επίσης η κατάσταση στο γάλα άλλαξε. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ε, αυτό, ε, αν γίνει διόρθωση πρέπει να αυξηθούν οι ποσοστώσεις σε μια ε, περίπτωση όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπερπροσφορά. Είναι λοιπόν αυτή η σωστή αντίδραση. Βλέπουμε ότι μειώνει η κατανάλωση του γάλακτος όπως και οι εξαγωγές του, άρα είναι η σωστή απόκριση να κάνουμε πιο ευέλικτους τους κανόνες για τις ποσοστώσεις το τελευταίο έτος. Τέταρτον, προκυπευτικά διάκριση μεταξύ οργανώσεων παραγωγών και παραγωγών που δεν είναι σε ενός παραγωγών. Ε, αυτή είναι μια στάνταρ πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομίζω υποστηρίζεται και από το κοινοβούλιο σας. Να υποστηρίξουμε δηλαδή, να ενισχύσουμε να τον ενισχύσω με τη θέση μεμονωμένων παραγωγών σε αυτό το τομέα ε, που ε, είναι έκθετη σε πιέσεις της αγοράς γιατί τώρα αυξάνει τη δυσκολία, έρχεται η συγκομιδή, πρέπει να τη διαθέσετε. Ο καλύτερος τρόπος, ε, θα συμφωνήσετε, είναι η οργάνωση των παραγωγών. Ένα παράδειγμα, αν εσείς ως μεμονωμένος παραγωγός οπωροκυπευτικών έχετε τη δύσκολη επιλογή να κάνετε, δηλαδή θα μαζέψω το προϊόν, θα προβώ στη συγκομιδή, χωρίς να ξέρω πού θα πουλήσω ή δεν θα το μαζέψω και θα το πάω για να καταστραφεί. θέλετε να ξέρετε τι θα κάνει ο ανταγωνιστής ή ο φίλος σας ή ο γειτονάς σας. Γιατί δεν θέλετε να αποφασίσετε να μην ε, μαζέψετε τα φρούτα και να δείτε μετά ότι κάποιος άλλος πουλάει τα χλάδια του στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό οι οργανώσεις παραγωγών είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό σε χώρες όπου είναι καλή οργάνωση ε, η απορρόφηση των πιέσεων γίνεται πιο ανώδυνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα για αυτούς που είναι ανεξάρτητοι, γιατί και στα νεκταρίνια και στα ροδάκινα ε, και σε άλλα προκυπευτικά υποστηρίζομαι πολύ και αυτούς που δεν είναι μέσα στις οργανώσεις. Αλλά υπάρχει διάκριση, υφίσταται, γιατί υπάρχει το κίνητρο. Όταν υπάρχει κρίση είναι πολύ σημαντικό να είστε μέσα σε μια οργάνωση. Ε, και τώρα, ε, με τη βοήθεια της Μονίκ Παριά, του συναδέλφου, ε, θα ήθελα να περάσω στο, στα εξωτερικά μέτρα. Προώθηση. 30 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν μέσα, εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, και τώρα γίνονται συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία όπου θα πρέπει να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, δεν μπορούμε μόνοι μας ένα προφανές πράγμα είναι το εξής και θα το δώσω με παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τώρα για την πρόθεση των εξαγωγών στη Ρωσία. Θα ρωτήσω με τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται εδώ αν θέλουν να τα διατηρήσουν αυτά τα προγράμματα ή αν θέλουν να προσανατολίσουν τα κονδύλια αυτά ε, αλλού, σε άλλες χώρες, όπως σε αυξανόμενες αγορές στην Ασία και αλλού επίσης. Ε, τώρα, φραγμή, ε, υγειονομικά, ε, προβλήματα με την Τουρκία, με άλλες χώρες. Εκεί υπάρχει δυνατότητα. Ε, επίσης ε, υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ε, χωρών που έχουν πληγεί. Έχουμε υποψήφιες χώρες και άλλες χώρες που μπορούν τώρα να ωφεληθούν από την ε, παράκληση του, των εξαγωγών προς τη Ρωσία. Για τον ΠΟΕ θέλω να πω ότι οι συνάδελφοί μας στην Γενική Διεύθυνση Εμπόριο και ο Επίτροπος Δεχούχτ εξετάζουν τις ε, δυνατότητες να ε, υπάρξει μια συζήτηση για αυτά τα μέτρα, αλλά δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υποδιευθυντά, ο κύριος Βοητσεχόφσκι. Μας έστειλε μια, ένα σχέδιο επιστολής σχετικά με την προφορική ερώτηση που θα απευθυνθεί στην Κομισιόν. Ορίστε. Η συζήτησή μας δείχνει ότι συμφωνούμε πως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε πολλούς τομείς, για πολλούς τομείς της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Σε μερικές χώρες υπάρχει μεγάλη κρίση και θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο και τους συναδέλφους να προβλέψουν στην ημερήσια διάταξη της επόμενης μας συνεδρίασης ή μάλλον στην επόμενη σύνοδο την προφορική ερώτηση με συζήτηση που προτείνω. Δηλαδή, ποια μέτρα έχουν ληφθεί και θα ληφθούν από την Κομισιόν για την αντιμετώπιση της κρίσης της ενωσιακής αγοράς που απορρέουν από τα ρωσικές απαγορεύσεις των εισαγωγών. Και δεύτερον, η Κομισιόν προτίθεται ή όχι να διευρύνει το, τα μέτρα που έχει ήδη λάβει για να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς. Αυτό το ερώτημα προτείνω να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Προφορικό, προφορική ερώτηση με συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κατανοώ, βλέπω ότι γενικά η Επιτροπή μας δέχεται αυτό το αίτημα και θα υποβληθεί η προφορική ερώτηση γραπτός στην επόμενη Ολομέλεια. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, τους εκπροσώπους της δηλαδή. Και λέω τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το 19. 19 για τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων είναι από τα σημαντικότερα θέματα της Επιτροπής μας. Το φθινόπωρο ε, τώρα δηλαδή θα γίνει αναθεώρηση του κανονισμού που θα αντικαταστήσει την, ε, το υπάρχον πλαίσιο με βάση τον κανονισμό 834 κάθετος 2007 με στόχο να αρθούν οι φραγμοί στην βιώσιμη παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ένωση να υπάρξει εγγύηση θεμητού και υγιούς ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τους εμπόρους και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Έμαθα ότι υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες της Κομισιόν σχετικά με αυτή την νομοθετική διαδικασία. Πρώτον, η Κομισιόν έχει προτείνει, εγκρίνει μάλλον ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής στην Ένωση. Δεύτερον, η Επιτροπή έχει πάρει εντολή από το Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών με βάση τις προτινόμενες αλλαγές σε αυτό το εμπορικό καθεστώς. Καλωσορίζω εδώ τον εκπρόσω... την εκπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Μονίκ Παριά, που θα παρουσιάσει την πρόταση και ζητώ περισσότερη πληροφόρηση για την εντολή των εμπορικών για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο τον Ιούνιο. Κυρία Παριά, έχετε τον λόγο. λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να υποφεληθώ με την ευκαιρία που μου δίνεται για να συγχαρώ τον εισηγητή που αν κατάλαβα καλά μόλις ορίστηκε υπεύθυνο για το θέμα αυτό Σας παρουσιάζω λοιπόν σήμερα την πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Βιολογική Γεωργία. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων αυξάνεται κατά 10% το χρόνο πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αντιπροσωπεύει και η Ένωση με τη ΣΥΠΑ μαζί αντιπροσωπεύουν το 90% της διεθνούς αγοράς βιολογικών προϊόντων που χωρίζεται μισό-μισό περίπου μεταξύ των δύο. Η βιολογική γεωργία καλύπτει 10 εκατομμύρια εκτάρια και είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι κατά μέσο όρο η βιολογική παραγωγή είναι νεότερη και οι περισσότερες γυναίκες. Είναι λοιπόν τομέας που δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει, αντιπροσωπεύει πολλά ωφέλη για την ε, ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στην Ένωση. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά είναι επίσης φανερό ότι ο τομέας αυτός διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί αρνητικές συνέπειες από την ίδια του την επιτυχία. Γι' αυτό αποφάσισε να αντιδράσει η Κομισιόν για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν είμαστε οι μόνοι που διαπιστώνουμε ότι η πολυπλοκότητα και το γραφειοκρατικό άχθος του καθεστώτος που επιβάλλεται στα βιολογικά προϊόντα είναι κάτι το απαράδεκτο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βιολογική παραγωγή αναπτύσσεται δύο φορές πιο αργά από ότι η αγορά των, εισαγωμένων προϊόντων. Οι μικρές, τα μικρά αγροκτήματα, κάτω από 5 εκτάρια δηλαδή, είναι τα περισσότερα από τα βιολογικά. Οι απάτες που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι έχει όρια το υπάρχον σύστημα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Εξάλλου το ελεκτικό συνέδριο έκανε ορισμένες συστάσεις με στόχο να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου που έχουμε. Δεν προβλέπεται καμία αμοιβαιότητα αυτή τη στιγμή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τα βιολογικά προϊόντα. Γι' αυτό αντιδράσαμε για να βρούμε λύσεις για τα αιτήματα αυτά του ελεγκτικού συνεδρίου ώστε να διασφαλίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των παραγωγών οι οποίοι πρέπει να μπορέσουν να υποφεληθούν από τις ευκαιρίες που μας δίνει η αγορά. Οι δε καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην βιολογική παραγωγή και στα βιολογικά προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν. η Κομισιόν άρχισε τη διαδικασία προετοιμασίας της διαρρύθμισης αυτής παραγγέλνοντας μία μελέτη αλλά επίσης, ε, όχι μόνο μεταξύ των εκπροσώπων του τομέα, αλλά και μεταξύ καταναλωτών, επιστημόνων, αγροτικών συμβουλίων, εκπροσώπων τρίτων χωρών, του ακαδημαϊκού κόσμου, του λιανικού εμπορίου, της μαζικής ε, εστίασης των προϊόντων δίκαιου εμπορίου κλπ. Προσπαθήσαμε, προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε μια πολύ ευρεία διαβούλευση για να καταλήξουμε σε μια πρόταση που να ανταποκρίνεται στις περισσότερες ευχές και ανησυχίες των κυρίων ενδιαφερομένων. Από αυτή τη δουλειά καταφέραμε να διατυπώσουμε διάφορα σενάρια των οποίων οι ποιοτικέ επιπτώσεις και οι ποσοτικές ε, περιγράφονται στην αξιολογική ανάλυση που συνοδεύει την παρουσίασή μας, την πρότασή μας. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν έτυχαν διαβούλευση σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, 1,5 χρόνο τώρα. Ιδιαίτερα η Κομισιόν άρχισε διαβούλευση για την αναθεώρηση που έλαβα, όπου έλαβαν χώρα 45.000 απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και φάνηκε ότι ενδιαφέρει τους πολίτες η βιολογική γεωργία. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες και την αξιολογική ανάλυση αποφασίσαμε λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση που έχετε τώρα μπροστά σας. Θα σας θυμίσω σύντομα τους κύριους στόχους της πρώτον να αρθούν οι φραγμοί για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ένωση, ιδιαίτερα να απλοποιηθούν και να ελευθερινθούν τα γραφειοκρατικά άχθη που αντιμετωπίζει. Από την άλλη να υπάρξει θεμητός ανταγωνισμός και καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων και τρίτον, το είπα λίγο και πριν, να εγγυηθούμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τα βιολογικά προϊόντα ότι δηλαδή τα βιολογικά προϊόντα που θα καταναλώνει παράγονται με βάση διαφανή και σαφή κριτήρια. Θέλουμε επίσης να υπάρχει η ίδια ποιότητα σε όλα τα ευρωπαϊκά βιολογικά προϊόντα με τα εισαγόμενα. Τέλος. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που έχουμε σαν στόχο επειδή έχει μεγάλο δυναμικό τομέας αυτός και δημιουργεί και θέσεις εργασίας να εγγυηθούμε και τη διεθνή του προβολή. Θα σας αναφέρω επίση γενικά τι λέει η πρόταση αυτή και ποιες προτάσεις περιέχει για να εφαρμοστούν οι στόχοι αυτοί. Προτείνουμε λοιπόν απλοποίηση της νομοθεσίας και μείωση του διοικητικού της κόστους. Η Κομισιόν απλοποίησε το υπάρχον κείμενο που ήταν αυτό δυνατόν για το εύρος εφαρμογής προβλέπουμε να μην παραπέμπουμε μόνο σε ορισμούς που χρειάζονται συνεχή αλλαγή αλλά σε έναν απλό κατάλογο προϊόντων των δύο συνημένων ή προστικών του κειμένου. Για το γραφειοκρατικό άχθος η πρόταση της Κομισιόν θα επιτρέψει τη μείωση κατά 25 περίπου της 100 το άχθος αυτό, μειώνοντας τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του άχθους για τις εθνικές, τα εθνικά υπουργεία. 37 λοιπόν τέτοιες υποχρεωτικές πληροφορήσεις θα καταργηθούν. Το πέρασμα από έναν έλεγχο βασιζόμενο στην ανάλυση του κινδύνου που να αντικαθιστά το υπάρχον σύστημα ετησίου ελέγχου θα συμβάλλει επίσης σε περισσότερη αποτελεσματικότητα και καταλληλότερη καλύτερη χρήση των πόρων. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικροπαραγωγών στην αγορά των βιολογικών προϊόντων όπως ζήτησαν ορισμένες οργανώσεις των μικροπαραγωγών, η εφαρμογή ενός συστήματος πιστοποίησης έχει προταθεί, το οποίο σύστημα ήδη χρησιμοποιείται από μερικές τρίτες χώρες και επιτρέπει σε μικροπαραγωγούς να εφαρμόσουν πιο εύκολα τον απαραίτητο έλεγχο και πιστοποίηση για να βελτιώσουν την εμπορία των προϊόντων τους. Για να υπάρξει θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών αυτών για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προτείνεται να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα, δηλαδή να καταργηθούν πολλές από τις υπάρχουσες εξαιρέσεις, πράγμα το οποίο ζήτησαν πολλοί καταναλωτές και πολίτες κατά τις διαβουλεύσεις μας, αλλά και ελεγκτές. Η κατάργηση των εξαιρέσεων θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και καταναλωτριών που θα έχουν την εγγύηση ότι θα αγοράζουν βιολογικό προϊόν ίδιας ποιότητας από όπου και αν προέρχεται. Η ενδυνάμωση, η ενίσχυση των ελέγχων θα αυξήσει επίσης την αποτελεσματικότητα μέσω της συγκέντρωσης της προσοχής στους τομείς όπου υπάρχουν οι έχουν διαπιστωθεί οι περισσότεροι κίνδυνοι και απάτες και όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας θα υποβάλλονται στους ελέγχους αυτούς καθώς και οι λιανοπολιτέ που αυτή τη στιγμή εξαιρούνται. Επίσης οι επόπτες, οι ελεγκτές μας ζήτησαν να καταργηθεί η εξαίρεση που προβλέπει ότι μία ολόκληρη σοδιά πρέπει να ελέγχεται βιολογικά. Γιατί είναι υπερβολικά μεγάλος ο κίνδυνος απατών εδώ η διεύρυνση της διεθνούς διάστασης της πολιτικής μας διασφαλίζεται μέσω των διατάξεων για τις εξαγωγές. Σε πνεύμα αμοιβαιότητας θα θέλαμε να βελτιωθεί η πρόσβαση βιολογικών προϊόντων και σε άλλες αγορές για να μπορούν οι ενωσιακοί παραγωγοί να υποφεληθούν από πιθανές αγορές εκτός Ένωσης. Μέχρι τώρα η πολιτική μας για τη βιολογική γεωργία δεν ασχολούνταν παρά μόνο με τη διευκόλυνση εισαγωγών από τρίτες χώρες. Θελήσαμε να προσθέσουμε και μία διάσταση προώθησης των εξαγωγών προς τρίτες χώρες. Όπως τονίσατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, μαζί με αυτές τις διατάξεις προτείνουμε και ένα σχέδιο δράσης για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων που αποτελεί την Ευρω... τη στρατηγική της Κομισιόν για την εφαρμογή, καλύτερη εφαρμογή αυτών των προτάσεων και την ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων στην Ένωση. Γνωρίζετε ότι οι προτάσεις αυτές είναι μία από τις δύο προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας με την οποία αρχίσαμε τις συνεννοήσεις πριν το καλοκαίρι, με το Συμβούλιο δηλαδή, και ήδη από την προηγούμενη ελληνική προεδρία. Η Κομισιόν χαίρεται ιδιαίτερα για την, πρόταση, για την πρόθεση αυτή της Ιταλικής Προεδρίας να γίνει σύντομη πρόοδος στο θέμα των βιολογικών προϊόντων για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως και ιδιαίτερα εδώ θέλω να επιμείνω, λόγω της δυνατότητας ανάπτυξης και απασχόλησης που αντιπροσωπεύει ο τομέας αυτός, όχι μόνο για την παραγωγή αλλά και για τη μεταποίηση και διανομή των προϊόντων αυτών. Χαίρομαι για τη συνεργασία μας για το ενδιαφέρον αυτό θέμα και προσδοκώ την συνέχεια της πολιτικής μας συζήτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ο κύριος Έριξον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα να πούν ότι ο κλάδος αυτός αναπτύσσεται και έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα σήμερα από ό,τι στο παρελθόν και δημιουργούνται όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα και φυσικά και εισόδημα για τους γεωργούς. Όμως υπάρχουν και προβλήματα με τον προτινόμενο κανονισμό. Αν και η βασική ιδέα είναι καλή, φαίνεται ότι δημιουργούν οι προτάσεις αυτές τώρα προβλήματα για πολλούς γεωργούς. Παίρνουν το σχάρι συνομιλώντας με τους Σουηδούς παραγωγούς και τις οργανώσεις παραγωγούν, μου είπαν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική μείωση της βιολογικής παραγωγής, ε, ίσως και κατά 80% αν τεθεί σε εφαρμογή, γιατί οι προτάσεις τους δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Δηλαδή για τις μικρές ομάδες, ε, για τους σπόρους πράγμα που πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να μεγεθυνθεί ο τομέα και να λειτουργεί καλά στο μέλλον. Χρειαζόμαστε αρκετέ αλλαγέ στις προτάσεις για να είναι καλή η νομοθεσία και θετική για τον κλάδο. Διαφορετικά, πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο πιστεύουν ότι καλύτερα είναι να συνεχίσουν με την ισχύουσα νομοθεσία παρά να έχουμε κάτι εντελώς καινούριο. Ευχαριστώ. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε σε διάφορες ε, περιπτώσεις. Ε, θα ήθελα να κρατήσετε το χρόνο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Αντρία. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν που μας παρουσίασε το πλαίσιο μέσα στο οποίο υποβάλλεται η πρόταση αυτή σήμερα. Το δικαίωμα είναι να επιτρέψουμε να μεγεθυνθεί αυτός ο τομέας και νομίζω ότι είναι μεγάλο διακύβευμα. Φυσικά ο στόχος ε, ε, είναι να τροποποιηθεί ο ισχύων κανονισμός και νομίζω ότι πρέπει να άρουμε τα εμπόδια στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά όμως υπάρχει και αναγκαιότητα να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ κρατών μελών. Όμως ε, είναι ουσιαστική και η διατήρηση κάποιας ευελιξίας για να ενθαρρύνουμε αυτό το τομέα να αναπτυχθεί και πιστεύω ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε και να επιτρέψουμε τόσο αυτή είναι η απόψή μου που συνάντησα ανθρώπους από τον κλάδο να προβλέψουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούν να υπάρχει διαχείριση της βιολογικής παραγωγής αλλά και της συμβατικής παραγωγής εντό της ίδιας εκμετάλλευσης. Το 23% των ε, εκμεταλλεύσεων σήμερα στη Γαλλία έχουν μεικτή παραγωγή. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να προσέξουμε τι θα υιοθετήσουμε Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητα για μικτές παραγωγές και εσείς το υπενθυμίσατε, θα πρέπει να οργανώσουμε αποτελεσματικά τους ελέγχους και θα πρέπει να υπάρχει ένα αρμονισμένος μηχανισμός μεταξύ των κρατών μελών. Εσείς ε, μας προτείνετε να προσφύγουμε μόνο σε ανάλυση κινδύνου. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια απέτηση που πρέπει να την αναλάβουμε οματικά. Κατάλαβα βέβαια από τις προτάσεις σας ε, ότι σε κάθε στάδιο της παραγωγής ε, υπάρχει αυτή η απέτηση για τον έλεγχο και συμφωνούμε. Και σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση που μας γίνεται, εγώ νομίζω ότι τίθεται και ένα ζήτημα επιτροπολογίας. Και πολλές από τις νομικές πτυχές που προτείνεται το κείμενο παραπέμπονται σε της πράξης. Εγώ νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να ενισχύσουμε τη βασική πράξη παρά να παραπέμπουμε αυτές τις νομοθετικά ζητήματα σε της πράξης. Αυτά ήθελα να πω για τη συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Ρεν. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι η αγορά βιολογικών προϊόντων αναπτύσσεται γρήγορα στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την σημερινή αλλά και τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Γεωργία. Επομένως είναι θετικό και η Κομισιόν και η Ιταλική Προεδρία έχουν θέσει αυτό το θέμα ως προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη βιολογική παραγωγή, αλλά ένα και περισσότερο. Από αυτή τη σκοπιά η σημερινή νομοθεσία για τα βιολογικά έχει λειτουργήσει καλά. Όμως δεν έχει απαντήσει σε όλες τις προκλήσεις της ε, βιολογικής παραγωγής, παραδείγματος χάρη. Αυτή είναι η περίπτωση στις πιο βαρύς ψυχρότερες συνθήκες. Και για στους λόγους αιτιολογείται η τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας και από τις αρχές την υποστηρίζουμε. Κάποιοι γεωργοί βιολογικών προϊόντων ε, ανησυχούν για κάποια από τα στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης. Η ανησυχία τους ήταν η κύρια ανησυχία τους ήταν ότι η μεταρρύθμιση θα καθιστούσε τη βιολογική γεωργία πιο δύσκολη από τη σήμερα. πρόταση Κομισιόν θα οδηγούσε σε περισσότερη γραφειοκρατία και σε περισσότερους ελέγχους. Φυσικά, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη βιολογική γεωργία. Όμως, κατά την άποψή μας, αν ε, αυξήσουμε του ελέγχου και την γραφειοκρατία, αυτό δεν θα οδηγήσει απαραίτητα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντίθετα, υποστηρίζουμε τη μετάβαση σε μία εποπτεία που θα βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων και θα είναι πιο αποτελεσματική. Όμως επί της αρχής ε, δεν απαιτούνται νέα αυξημένη έλεγχη στο βιανικό εμπόριο, την χάρη για τα βιολογικά προϊόντα. Αντίθετα, θα πρέπει να στοχεύουμε στο να μειώσουμε την γραφειοκρατία που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε κρόμιση κόστου και στο πλαίσιο αυτό η γεωργοί μικρή κλίμακα θα πρέπει ιδιαίτερα να ληφθούν υπόψη. Συνολικά, η Κομισιόν κάνει μια πρόταση που χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις και αλλαγές πριν να μπορεί να τεθεί σε ισχύ. Παραδείγματο χάρη, αυτό αφορά την απέτηση να ε, αλλάχθεί όλη η παραγωγή της εκμετάλλευσης και να μεταμορφωθεί σε βιολογική παραγωγή. Πάντως θεωρούμε ότι η σημερινή πρόταση είναι σημαντικά βελτιωμένη. Ευχαριστώ κυρία Σχάιερ. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιεί τη βιολογική γεωργία τώρα, αλλά δεν υπάρχει ενιαίο μέτρο σύγκριση των εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ευρώπη. Στη Φιλανδία, στην Ελλάδα, στην Ολλανδία εργάζονται διαφορετικά. Αν τυποποιήσουμε τις διαδικασίες, δεν θα έχουμε ίσους όρους του παιχνιδιού, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και οι αγρότες και οι αγρότησες ε, θα πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές. Ε, μιλάμε για τη βιολογική γεωργία. Ο κανόνας είναι η διαδικασία παραγωγής να είναι απόλυτα βιολογική και για ορισμένες επιχειρήσεις αυτό απλώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Ε, δεν υπάρχουν αυτές οι δεξιότητες. Πρέπει λοιπόν να δουλεύει η Κομισιόν με πιο ευέλικτους ορισμούς της βιολογικής γεωργίας που θα μας εξυπηρετεί θα μας εξυπηρετούν περισσότερο. Ας πούμε υπάρχουν μικτάες εκμεταλλεύσεις ε, πολλές φορές που πρέπει να καλύπτονται. Δεν μπορούμε πολλές φορές να ε, έχουμε 100% ε, βιολογικά προϊόντα. Μπορούμε να έχουμε εν μέρη. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπή, συνάδελφοι, με την πρόταση αυτή της Κομισιόν έχουμε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό. Και αν μετρήσω την Κομισιόν με βάση αυτά που είπε και ε, που αποσκοπεί, όπως είπε, με την πρότασή της να μειώσει την γραφειοκρατία και να επεκτείνει την βιολογική γεωργία, πρέπει να πω ότι από πολλές συζητήσεις ε, με τους ε, εμπλεκόμενους. Ε, μπορώ να πω ότι με πολύ επικριτικό μάτι αντιμετωπίζεται την πρόταση που δεν θα μειώσει όπως θεωρούν τη γραφειοκρατία εκτός από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχει και πολλά σημεία που καλύπτονται με κατεξουσιοδότηση πράξης με τις οποίες έχουμε πολλά προβλήματα. Αυτό το σύστημα δηλαδή γίνεται αμφισβητήσιμο με τις πράξεις αυτές. Η Κομισιόν δεν πρέπει να κάνει ως εάν τώρα ανακάλυψε τη σημασία του τομέα, το εξαγωγικό του δυναμικό κλπ. Οι, βιο, ενώσεις βιολογικών ε, προϊόντων ε, από μόνες τους εξελίχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ε, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πλήρες κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό. Καταρχήν ε, είχαν γίνει κάποιες, ε, είχε, γίνει ένα ερωτηματολόγιο που και αυτό ήταν προβληματικό γιατί ήταν ασαφείς οι ερωτήσεις και τα αποτελέσματα δεν θα ήταν αξιόπιστα ή θα ήταν αυτά που ήθελε η Κομισιόν. Δηλαδή ε, αν ε, ε, παράγουν προϊόντα ε, τα χωρίς ευλαβερές ουσίες εκεί όλοι θα απαντήσουν ναι. Στα κατάλοιπα υπάρχουν κάποιες οριακές τιμές που προσανατολίζονται σε κάποιες σταθερές. Αυτό είναι καλό. Ε, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας πού ε, ασκείται η βιολογική γεωργία, σε ένα περιβάλλον εμπορικής γεωργίας και δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε υπεύθυνου ε, αν ε, ορισμένα προϊόντα έχουν ένα ποσοστό για παράδειγμα ζυζανιοκτώνων τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι αλλά ε, προέρχονται από τους γείτονες, από γειτονικέ καλλιέργειες. Ε, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, το μέλλον θα δείξει συνέχεια. αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα γιατί συνεπάγεται ε, πολλά νομικά θέματα, νομοθετικά θέματα, τα οποία δημιουργούν μάλλον ανησυχία και αβεβαιότητα στους βιολογικούς ε, παραγωγούς παρά τους καθησυχάζουν. Ε, ε ο πρόεδρος μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσω για να ολοκληρώσω. Πώς αντιμετωπίζουμε τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων. Ε, υπάρχουν εδώ εμπορικές συζητήσεις και, που θα οδηγήσουν σε συμφωνίες πλαίσιο ε, το πρόβλημα δεν εξαντλείται όμως εκεί. Ιδιαίτερα οι εισαγωγές είναι ένα τεράστιο θέμα και θα πρέπει να βρεθούν ρυθμίσεις που στο μέλλον θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε αμοιβαία, ρύθμιση, αμοιβαία αναγνώριση πάντα των προτύπων των άλλων χωρών και να αφήσουμε το θέμα εκεί. Όχι. Θα πρέπει να βρεθούν και άλλα κριτήρια. Αλλιώς ε, θα συρρυκνώσουμε τον τομέα αντί να τον διευρύνουμε. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για βιολογική παραγωγή, θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το δρόμο. Δηλαδή να χρησιμοποιούν 100% οικολογικό σπόρο. Αυτό το δεχόμαστε και το θέλουμε όλοι. Πρέπει όμως να έχουμε την αγορά για οικολογικούς σπόρους. Δεν μπορώ να ζητήσω 100% να έχει οικολογικό ε, σπόρο όταν δεν μπορεί να τον βρει τον σπόρο αυτό. Πρέπει να τον διευκολύνουμε για να το κάνει αυτό. Ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη, τα καινούρια που δεν υπάρχουν τέτοιες αναπτυγμένες δομές. Πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες ε, εξαίρεσης, ούτως ώστε να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή και να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την ολοκλήρωση του τομέα της βιολογικής γεωργίας. Ε, δεν μπορούμε εν μια νυχτή να τα κάνουμε όλα, διότι θα φοβηθούν οι γεωργοί και δεν θα κάνουν τη μετάβαση στη βιολογική γεωργία. Θα θεωρήσουν ότι είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ο κίνδυνος αν δεν τα διευκρινίσουμε αυτά, μπορεί να μειωθεί η βιολογική καλλιέργεια αντί να αυξηθεί. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα επιτύχουμε αυτό τον απότερο στόχο μας. Να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των ε, παραγωγών και να αυξήσουμε τη βιολογική γεωργία. ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν να πω ότι με ανησυχεί η υπερβολική ανησυχία της Κομισιόν για τον εξαγωγικό προσανατολισμό για τα βιολογικά προϊόντα και με ανησυχεί γιατί όταν κάτι τέτοιο θέλουμε να ενισχύσουμε τελικά γίνεται πολύ μεγάλη επίθεση στην αγροτιά και υπάρχει εξάρτηση από τις πολυεθνικές αν αναφέρω το παράδειγμα των σπόρων, στο οποίο αναφέρθηκε και ο προηγούμενος ομιλητής, αν ε, εδώ ε, τελικά καταλήξουμε να μην έχουμε τοπικούς σπόρους, τότε οι γεωργοί θα εξαρτώνται πάρα πολύ από τις πολυεθνικές για τους σπόρους. Και το δεύτερο που θέλω να θέσω στην Κομισιόν, αν μπορεί να θεωρηθεί οικολογικό, ένα βιολογικό προϊόν που θα μπορούσε να παραχθεί σε κάθε μία από τις χώρες μας, και ε, τελικά το καταναλώνουμε αφού έχει εξοδευτεί πάρα πολύ ενέργεια και έχει διατρέξει πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Μπλάνεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Απλά ήθελα και εγώ να φερθώ στο είπαν συνάδελφοι για την προτείνομενη απαγόρευση για παράλληλη βιολογική ε, και συμβατική παραγωγή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 20% από τους αγρότες προβαίνουν και σε συμβατική παραγωγή, ίσως γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη αγορά για τα βιολογικά προϊόντα για να έχουν 100% βιολογική παραγωγή και επίσης πολλοί βρίσκονται σε κάποια μετάβαση από τη συμβατική στη βιολογική παραγωγή. Δεν μπορεί να γίνει εν μία ανοιχτή και αν ακολουθήσουμε αυτή την οδό και απαγορεύσουμε την παραγωγή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διαστρεβλωμένο ε, μια δεστρεμμένη συνέπεια να σπρώξουμε τους γεωργούς πάλι πίσω στη συμβατική γεωργία και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ εκτιμώ την πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή και είναι απαραίτητη. Διαφωνώ με κάποιους από τους προηγούμενους ομιλητές σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των συνθήκων για τη βιολογική γεωργία, για τα βιολογικά προϊόντα. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και κάθε γεωγραφικής περιοχής. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δεκτούμε ότι ένα προϊόν που παραδείγματος χάρη έρχεται από τη Ρουμανία μπορεί να έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αζωτούχων από ένα προϊόν από την Ιταλία, ή τη Γερμανία παραδείγματο χάρη. Χρειαζόμαστε ένα βαθμό τυποποίηση ε, των κριτηρίων προκειμένου να δηλώσουμε στη Γεωργία ότι έχουμε βιολογικό προϊόν. Όμω από την άλλη πρέπει να μειώσουμε και τη γραφειοκρατία. Γιατί η γραφειοκρατία απλώ αποθαρρύνει του ανθρώπου από το να περάσουν στη βιολογική γεωργία και νομίζω ότι χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερου βιολογικού γεωργού που μπορούμε να έχουμε. Σα ευχαριστώ. Κυρία Χέρανς Γκαρσία είναι τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία του Βρετανού συναδέλφου Νομίζω ότι ενώ γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η βιολογική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η πρόταση να εξελιχθούν οι μεικτέ εκμεταλλεύσει μπορεί να επιφέρει σημαντικού κινδύνου για την ίδια τη βιολογική παραγωγή. Ενώ αυξάνεται η ζήτηση, δεν φαίνεται λογικό να βάλουμε σε μια βολή θέση του παραγωγού οικολογική γεωργία ε, που έχουν παράλληλη παραγωγή για να του κάνουμε ε, να επιλέξουν, γιατί είναι πολύ πιο ακριβή η βιολογική παραγωγή από τη συμβατική και τελικά θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή θα εγκαταλείψουν τη βιολογική παραγωγή γεωργή για να ξεκινήσουν συμβατική παραγωγή. Εγώ νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και να εργαστούμε κομισιόν για να τροποποιήσουμε την πρότασή της. Επίσης, για τις ε, εξαιρέσεις πρέπει να τις σκεφτούμε λίγο περισσότερο αυτό το κεφάλαιο εγώ θα το εξετάζα πολύ προσεκτικά γιατί νομίζω ότι μπορεί σε ορισμένες ε, περιοχές όπου έχουμε σημαντική βιολογική παραγωγή να δημιουργήσουμε κάποια ζητήματα. Στο 40% των εκμεταλλεύσεων στην Ισπανία είναι μικτές και ποτέ δεν υπήρχε καμία περίπτωση απάτης. Αν δηλαδή υπάρξει κάποια απάτη πρέπει να αυξήσουμε τους ελέγχους, όλο και να εξελίψουμε τις εκμεταλλεύσεις και χρειάζονται και εξαιρέσει ε, στην Ισπανία για να μπορούμε να συνεχίσουμε με τη βιολογική γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Παριά σύντομα παρακαλώ. Θα υπάρξει έκθεση και θα επανέλθουμε, θα καταρτήσουμε έκθεση και θα επανέλθουμε στο θέμα. Έχετε το λόγο. Πανή Δρέκτορ Sorry, pardon, excusez-moi, mais j'avais plus Με συγχωρείτε, δεν ακούγα τη διερμηνία. Σας ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία για να ξαναδοθούμε. Βέβαια υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία προκάλεσαν αντιδράσεις ε, από την πλευρά σας. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω τα σχόλιά σας. Γραφειοκρατία. Είναι σαφές ε, και το είπα στις αγωγικές μου παρατηρήσεις ότι ένας από τους στόχους αυτής της μεταρρύθμισης είναι να μειώσει το, το δικαιωτικό κόστος και τη γραφειοκρατία. Καταθέσαμε μια πρόταση η οποία είναι βελτιώσιμη βεβαίως, αλλά είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους που έχουμε στη μεταρρύθμιση, δηλαδή να μειώσουμε το δικαιωτικό κόστος και την γραφειοκρατία. Οι προτάσεις σας λοιπόν για τη βελτίωση της πρότασης είναι καλοδεχούμενες και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σας. Εκτιμούμε ότι η πρόταση που έχουμε καταθέσει ήδη μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της γραφειοκρατίας, ιδίως μειώνοντας τον αριθμό των εξαιρέσεων, μειώνοντας τις, μειώσεις, τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και επικεντρώνοντας τους ελέγχους στους πιο επικίνδυνους τομείς ή στις πιο επικίνδυνες εκμεταλλεύσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αντίκτυπο που θα είχε η πρόταση αυτή επί του επιζητούμενου στόχου. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αποφύγουμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της εμπιστοσύνης που θα πρέπει να έχουν οι καταναλωτές στο βιολογικό λογότυπο Όλοι είμαστε καταναλωτές όταν αγοράζουμε ένα προϊόν που έχει μια βιολογική ετικέτα. Πίσω από αυτό κρύβονται κάποιοι κανόνες, ε, κάποιοι τρόποι παραγωγής που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Το πρόβλημα της σημερινής νομοθεσίας είναι ότι έχει πάρα πολλές εξαιρέσεις που ανοίγουν την πόρτα σε τρόπους παραγωγής που θα μπορούσαν να διαφοροποιούνται τα μάλλον ένας από τον άλλο και τελικά θολώνουν το τοπίο που μπορεί να έχει ο καταναλωτής ε, για το βιολογικό προϊόν που καταναλώνει. Και εκεί μπορούμε να έχουμε και ένα διαστρεβλωμένο αποτέλεσμα, δηλαδή να απομακρυνθεί ο καταναλωτής από το προϊόν γιατί δεν το εμπιστεύεται. Από την άλλη ούτε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ριζοσπαστικοί γιατί τελικά και αυτό θα αποθάρρυνε τον παραγωγό να επιδοθεί στη βιολογική γεωργία προσπαθήσαμε να καταθέσουμε μία πρόταση που επιχειρεί να βρει την ορθή ισορροπία, δηλαδή αφενός να επιτρέψει να υπάρχει αρκετή ευελιξία και έχουμε προβλέψει και μεταβατικές περιόδους, μεταβατική περίοδο και μπορούμε να τη συζητήσουμε από κοινού στην πρόταση της καταξιδότητας πράξης για τα μέτρα που θα ληφθούν για την μεταβατική περίοδο αλλά είναι προφανές ότι οι εξαιρέσεις, ο αριθμός των εξαιρέσεων που υπάρχει σήμερα, το μόνο που κάνει είναι να θελώνει την εικόνα των βιολογικών προϊόντων στα μάτια του καταναλωτή. Το πρόβλημα των ελέγχων αναφέρθηκε από ορισμένους από εσά. Και εδώ οι εκμεταλλεύσεις είναι αντικείμενο συστηματικών ετησίων ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται και σε ιδιαίτερα αξιόπιστες εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε εκμεταλλεύσεις που θέτουν κάποιο κίνδυνο. Το κόστος του ελέγχου είναι υψηλό, είναι μεγάλο άχθος για τις επιχειρήσεις ε, και για τους ελεγκτικούς οργανισμούς, αλλά ακόμη και για τους φορολογουμένους. Πιστεύω πως σε πολλούς τομείς μια ανάλυση κινδύνου είναι μια καλή προσέγγιση. Στο βαθμό που θα μας επιτρέψει αυτοί που συμπεριφέρονται σωστά να μειώσουν το κόστος, δηλαδή να αποζημιωθούν από τις προσπάθειες που κάνουν και να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν σε αυτή την οδό και να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες αλλά και το κόστος για τους ελέγχους στις εκμεταλλεύσεις που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Νομίζω ότι η λογική είναι σωστή, μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση, αλλά νομίζω ότι η λογική είναι καλή, δηλαδή να θέλουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Μια προσέγγιση η οποία ακολουθείται και στα περισσότερα συστήματα ελέγχου, είτε πρόκειται για χρηματοκορμικού ελέγχους ή άλλους, έτσι ώστε να έχουμε εξορθολογισμό του κόστους των ελέγχων και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Τώρα, το πρόβλημα των μεικτών εκμεταλλεύσεων. Σήμερα η βιολογική γεωργία μπορεί να συνεπάρχει με τη συμβατική. Εκτιμούμε ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει μακροπρόθεσμα να εξελιχθεί για τον εξή λόγο. Καταρχήν, κάποια προβλήματα εμπιστοσύνη υπάρχουν σε ό,τι αφορά την παραγωγή, γιατί το είπατε κι εσεί. Είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε ότι κάποιε ουσίε που χρησιμοποιούνται συμβατική γεωργία δεν διαρέουν στο αγροτεμάχιο της βιολογική γεωργίας. Από την άλλη, ο κίνδυνος της απάτης είναι πιο υψηλός όταν ένα ε, πάει και επιτόπου και βλέπει σακιά με φυτοφάρμακα που δεν χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία και χρησιμοποιούνται την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να κάνει τη διάκριση μεταξύ των δύο εκμεταλλεύσεων και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει απάτη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλό αυτό, αλλά θα πρέπει να προβλέψουμε και μεταβατικές περιόδους για τους σπόρους. Να επενθυμίσω ότι για τους σπόρους έχουμε προβλέψει μεταβατική περίοδο για τη χρήση των σπόρων και των αναπαραγωγικών ζώων μέχρι το 2021 έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτρέψουμε τη χρήση των σπόρων καθαρά βιολογικού χαρακτήρα. Για την επιτροπολογία, όντως παραμπέμπουμε σε πολλές κατεξουσιοδότηση πράξεις και σε εκτελεστικά μέτρα. Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας να έχουμε πολύ σαφείς κανόνες και της αναγκαιότητας να μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες ανάλογα με την εξέλιξη της βιολογικής παραγωγής και της, βιολογικής, ε, και της τεχνολογικής έρευνας στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. θα ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, αλλά θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Όπως είπε και ο κύριος Ρεν, η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες. Πάμε στο επόμενο σημείο. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Οι γραμματείς, οι, πεταμέλη, η γραμματεία, οι πολιτικοί σύμβουλοι θα παραμείνουν στην αίθουσα. Διακόπτουμε για μισό λεπτό για να κάνουμε τα δέοντα και αρχίζουμε πάρα αυτά. Ευχαριστώ.